Καλή σας ημέρα. Καλωσορίζω θερμά όλους όσους καταφέρατε να φτάσετε σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Μεταδίδεται όπως πάντα στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μας. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι η ομάδα των περασίνων. Τη στήριξαν βέβαια και οι σοσιαλιστές και το ΕΛΚ. Ζήτησε αλλαγή της μερίσιας διάταξης. Δηλαδή, η ψηφοφορία να λάβει χώρα όχι το προέλατο απόγευμα, ώστε να έχουν καταφέρει να έρθουν περισσότεροι συνάδελφοι στις Βρυξέλλες. Αν λοιπόν δεν έχετε αντίρρηση και συμφωνείτε, θα μεταφέρουμε τις ψηφοφορίες το απόγευμα στις 4 και μισή, αμέσως μετά από την ακρόαση δηλαδή που έχουμε μαζί με την Επιτροπή Ήτρε. Αντί να ψηφίσουμε λοιπόν στις 10.30 το πρωί, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας για το γενικό κανονισμό. Το σημείο 12 δηλαδή, το σχέδιο μερικής διάταξης. So if there is no opposition to this... Αν λοιπόν δεν υπάρχει αντίρρηση προς την αλλαγή αυτή στην μερική διάταξη, την τροποποιούμε Όπω σα προανέφερα και περνάμε στο σημείο 2. Ανακοινώσει τη Πρόεδρου δεν υπάρχουν μέχρι στιγμή ανακοινώσει. Άρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 τη σημερινή διάταξη. Το σημείο του Γιάνν Όλμπριχτ. Εξέταση του σχεδίου έκθεση του κ. Όλμπριχτ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξη. Να σα υπενθυμίσω ότι στην Επιτροπή τη Συνεδρίαση στη τη επιτροπής μας στις 8 ε, του μήνα είχαμε συμφωνήσει ότι την 31η Μαΐου και 6 ώρα το απόγευμα θα λήξει προθεσμία την κατάσταση τροπολογιών. Κάτι άλλο που μπορεί να γνωρίζετε, θα σας το πω όμως, είναι ότι έχει μεταφραστεί έκθεση σε όλες τις γλώσσες. Είναι έτοιμη η μεταφράση ήδη από τις 24 Μαΐου. Για να έχει το λόγο, έχουμε χρόνο μέχρι τις 9.40 για την εκθεσή σου. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά γιατί είχα προετοιμάσει το κείμενο στα αγγλικά. Ξέρω ότι είναι μεταφράσει Έχουν διανεμηθεί σήμερα το πρωί μάλιστα. Έτσι ενημερώθηκα. Και να ξέρετε, συνάδελφοι, όσοι θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες μέχρι αύριο ότι υπάρχουν οι μεταφράσεις να σας αναφέρω τις προτάσεις μας. Ουσιαστικά μια πρόταση, μια σειρά τροπολογιών στην πρόταση της Κομισιόν. Αυτό που είναι σημαντικό καταρχάς ε, είναι ο κανονισμός για το ταμείο αυτό. Τι μορφή θα έχει. Επηρεάζεται από το λεγόμενο γενικό κανονισμό. Δηλαδή, τα βασικά στοιχεία περιλαμβάνονται στο γενικό κανονισμό και το Ταμείο είναι η συνέπεια της απόφασης που θα λάβουμε για το γενικό κανονισμό. Σε ό,τι αφορά τώρα τους θεματικούς στόχους, τη θεματική συγκέντρωση, thematic concentration, που είναι η βάση, οι επιπτώσεις δηλαδή του Ταμείου αυτού αλλά και του Κοινωνικού Ταμείου. Και το επόμενο είναι ο προγραμματισμός. Στο Γενικό Κανονισμό έχουμε τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, που έχει επιπτώσεις βέβαια για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα των χρηματοδοτικών μέσων, που και αυτά είναι στον γενικό. Νομίζω λοιπόν ότι στην ε, διάρκεια της τρέχουσας περίοδου προγραμματισμού θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και θα πρέπει να αναλύσουμε ταυτόχρονα τους κανονισμούς όλου συγχρόνω για να δούμε κατά πόσον είναι συμπληρωματικοί μεταξύ του. Γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν αντιφάσει μεταξύ των διαφορετικών κανονισμών και των διαφορετικών ταμείων. Εξίσου σημαντικό για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι το πρόβλημα του CSF και των κονδυλίων του. Κάποια από τα στοιχεία του CSF επηρεάζουν και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα πρέπει να δούμε τι τελική μορφή θα λάβει ο σχετικός κανονισμός. Τελευταίο σχόλιο για τον γενικό κανονισμό. Σχέση μεταξύ RDF-ESF, Κοινωνικού Ταμείου Περιφερειακού Ταμείου, Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει να κάνει και με τη χρηματοδότηση. Ένα σημαντικό επίστοιχο για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι οι προτινόμενες μέθοδοι για τη νέα περίοδο προγραμματισμού και συγκεκριμένα το ITI που ναι μεν είναι στον γενικό κανονισμό αλλά ε, επηρεάζει και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ό,τι αφορά τώρα τη δική μου πρόταση. Σε ό,τι αφορά πρώτον τα καθήκοντα του Ταμείου, προτείνω να περιληφθεί η παράμετρος των δημογραφικών προκλήσεων στα καθήκοντα του Τάμιου. Σε ό,τι το άρθρο 3. Πεδίο ή εύρος στήριξης, scope of support στα αγγλικά. Υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία, αλλά και επίμαχα Δεν θέλω να μιλήσω αναλυτικά για τι αιτιολογικέ σκέψεις. Βλέπετε βέβαια ότι υπάρχουν στην εκθεσή μου τροπολογίες για τις αιτιολογικέ σκέψεις, ιδίως ό,τι αφορά τις τεχνολογίες των επικοινωνιών και πληροφοριών, τη σχέση με το ορίζοντα 2020, οι δείκτες κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν τα επόμενα βήματα, αν θέλετε, και τα επόμενα σκέλη του κανονισμού. Στο άρθρο 2 προτείνω να περιληφθούν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις και αδυναμίες. Λέω να περιληφθεί αυτό στα καθήκοντα. Σε ό,τι αφορά τώρα το scope of support. Είπαμε εδώ υπάρχουν κάποια επίμαχα, κροσεπίμαχα σημεία. Προτείνω να διευρυνθεί το πεδίο τα με Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό θα μπορούσε βέβαια να ε, εννοηθεί και ως διαγραφή της θεματικής συγκέντρωσης, δηλαδή η διάχυση αυτής της ε, συγκέντρωσης. Δεν έχω ακριβώς αυτό το στόχο. Θέλω να διατηρηθεί η θεματική συγκέντρωση, αλλά να είναι πιο ευέλικτη. Οι τελική δικαιούχοι, πρώτα βέβαια τα κράτη-μέλη, αλλά και οι τελικοί δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τους πραγματικούς στόχους που θέλουν να επιτευχθούν. Αυτό που προτείνω, για παράδειγμα, είναι οι λεγόμενες productive investments, παραγωγικές επενδύσεις, να επεκταθεί το πεδίο. Η Κομισιόν περιορίζει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ προτείνω να διευρυνθεί το πεδίο και να πούμε ότι ειδικότερα ΜΜΕ, in particular SMEs, να μην εξαιρεθούν όμως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και αυτό γιατί πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στους φορείς εκείνους που μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Για μένα λοιπόν είναι πολύ σημαντικότερες οι νέες θέσεις εργασίας και όχι το ποιο τις δημιουργεί. Αν μπορούν να τις δημιουργήσουν ε, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ε, ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή πιο πολύ με ενδιαφέρει ο στόχος, ο σκοπός και όχι τόσο ποιος θα τον επιτύχει αν οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν αισθέσεις εργασίες, θα πρέπει να μπορούν να το κάνουν αυτό. Βέβαια, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι όμως μόνο αυτές. Υποδομές επίσης, πολιτισμό και αθλητισμό. Εδώ τι βλέπουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε κοινωνικά, εκπαιδευτικά θέματα και θέματα υγείας. Αν όμως δούμε τι θα πει σημαίνει κοινωνικό σε γενικότερο και ευρύτερο επίπεδο, σημαίνει μεταφορές, πολιτισμό, υγεία, τα πάντα. Αν όμως η Κομισιόν προτείνει κοινωνικό, μετά λέει εκπαίδευση και μετά υγεία, άρα αλλιώς αντιλαμβάνονται την έννοια κοινωνικό. μάλλον κοινωνική πρόνοια, social care, education, health. Αν προτείνει αυτά η Κομισιόν, νομίζω ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλες υποδομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολιτισμός, επαναλαμβάνω, αθλητισμός και τουρισμός. Ο τουρισμός, να σας υπενθυμίσω, ότι είναι ένα από τα σημαντικά ε, στοιχεία της οικονομίας. Συνεδριάσαμε για τον τουρισμό στην ομάδα μας, στο ΕΛΚ, και δεν μιλάω για τον ελεύθερο χρόνο, μιλάω και για τη σημασία του τουρισμού στην οικονομία. Θα προτείνω επίσης στο άρθρο 3 συγκεκριμένα τα σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα διάφορες μορφές ε, παροχής βοήθειας, εγγυήσεις, δάνεια, μετοχές κτλ. Μιλάω επίσης για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, γιατί συζητάμε για ε, φορείς, όχι για πληθυσμό αν πούμε regions, towns, πόλεις, περιφέρειες, μιλάμε για όλον τον ε, πληθυσμό. Αλλά αν μιλάμε για τοπικές περιφερειακές αρχές, τότε μιλάμε ουσιαστικά για τους ενεργούς φορείς, για τους παράγοντες. Και το πρόβλημα των υποδομών, ε, άκρος επίμαχο και αυτό, θα πρέπει να επιτρέψουμε στις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες να επενδύσουν στην υποδομή για βασικές υπηρεσίες, στις μεταφορές, στο περιβάλλον και στις τεχνολογίες πληροφοριών επικοινωνιών. Μετά από συνεδριάσεις με πολλούς φορείς προτείνω διαγραφή. Δηλαδή να μην απαγορεύουμε στις πλέον ανεπτυγμένες περιφέρειες να επενδύουν σε υποδομές. Βρισκόμαστε σε καιρό κρίσης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπό αυτές τις συνθήκες η επένδυση σε αυτούς τους τομείς, στις υποδομές τομείς αυτούς είναι κατά της θεματικής συγκέντρωσης, όλο, ε, κάθε άλλο μάλιστα. αν είναι απαραίτητη θεματική συγκέντρωση για τη δημιουργία υποδομών, να είναι επιλέξιμη. Μπορούμε να πούμε όμως όχι βασικές υποδομές ε, ή τεχνολογίες πληροφοριών επικοινωνιών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 4, θεματική συγκέντρωση, ουσιαστικά πρόκειται για διαφορετικούς τρόπους ε, δημιουργίας μεγαλυτερη ευελιξια ε, Τρία στοιχεία περιέχει η πρότασή μου. Πρώτον να αλλάξουμε τους αριθμούς από το 8 να πάμε στο 7, από το 40 στο 30. Τρεις θεματικοί στόχοι. Έπειτα για τον τέταρτο θεματικό στόχο, δηλαδή ICT, τεχνολογίες προφόρων επικοινωνιών, να είμαστε πιο ευέλικτοι, να διευρύνουμε το πεδίο. Τέσσερις προτεραιότητες, ε, μάλλον για διάφορες προτεραιότητες όπως είναι η δαφική συνεργασία. Εδώ δεν έχουμε συμπληρωματικότητα. Και το τρίτο στοιχείο για την ενεργειακή απόδοση το ε, κατώτατο απαιτούμενο επίπεδο, εγώ λέω να, μειώσουμε εδώ τα νούμερα. Και ξέχασα και κάτι ε, στο άρθρο 3, τον καπνό συγκεκριμένα. Μέχρι τώρα, κανείς δεν μπόρεσε να με εξηγήσει γιατί κάτι το οποίο εντάσσεται στη Γενική Ευρωπαϊκή Πολιτική, κατά δηλαδή του καπνίσματος που συμφωνώ εγώ. Γιατί περιλαμβάνεται εδώ στο Ταμείο. Εγώ δεν λέω, ναι, δεν είμαι αντίθετο, αλλά γιατί περιλαμβάνεται εδώ. Απλά δεν βρίσκεται σωστό σημείο. Δεν λέω ότι είναι κακό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ε, προτεραιότητε στον τομέα των επενδύσεων. Βλέπω από το Συμβούλιο ότι ενώ μεν παραμένουν ε, τα κουτιά, διευρύνουμε το περιεχόμενο. Αυτό τι σημαίνει, είναι ενδιαφέρον. Επισήμως υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση, ανεπισήμως όμως όχι, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Όλοι κάτι προσθέτουν δηλαδή στις προτεραιότητες, άρα θα προσθέσω κι εγώ. Προτείνω λοιπόν καταρχάς, και αυτό όχι γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια σαφή, μια θολή εικόνα για την ε, θεματική συγκέντρωση, αλλά γιατί πρέπει να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Το συνέργειε με τον ορίζοντα 2020. Θα πρέπει να ανοιχτεί ανοιχτή η πόρτα για τη δημιουργία συνδέσεων με τον ορίζοντα 2020. Έπειτα το στοιχείο ε, των δημιουργικών βιομηχανιών, πολιτισμού. Άμεσα συνδεδεμένο σήμερα για μένα με την καινοτομία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θέλω να περιλάβουμε εδώ. Ανεξαρτήτως μεγέθους λοιπόν να περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις, τα ίδια με πριν, έπειτα συστήματα μεταφορών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και όπως με τις νέες θέσεις εργασίας που είχα πει. Τι μας ενδιαφέρει τελικά, να έχουμε χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Αν μας ενδιαφέρει αυτό θα πρέπει να είναι στη θεματική συγκέντρωση μεταφορές Περί αυτού πρόκειται. Αφού περί αυτού πρόκειται, πρέπει να μπει στη θεματική συγκέντρωση ο τομέα. Γι' αυτό προτείνω τη σχετική αλλαγή. Επίση, επενδύσεις σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ταστάσει ε, αποθήκευσης, βελτίωση αστικού περιβάλλοντος, αποκατάσταση σιδηροδρόμου, μεταφορά νερού κτλ. Πιστεύω μετά από πολλές συναντήσεις που έχω ότι αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να προσθεθούν και κατά την άποψή μου δεν μεταβάλλουν το περιεχόμενο των προτεραιοτήτων επενδύσεων. Μετά από πάρα πολλές συζητήσεις προτείνω επίσης διαγραφή των δικτών από το παράρτημα του κανονισμού. Είναι οι δείκτες παραγωγής output indicators που ουσιαστικά είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης δεδομένων και θα πρέπει να είναι σε κατεξουσιοδότηση πράξη και όχι στο ταμείο για τη βιώσιμαστική ανάπτυξη. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Στηρίζω το να έχουμε ένα 5% εθνικής κατανομής, αλλά αυτό να πάει στις λειτουργικές αστικές περιοχές, που θα ορίζονται στο πλαίσιο των συμβάσεων εταιρικής σχέσης. να καθορίσουμε κάποια κριτήρια και να δημιουργήσουμε και κάποια πιλωτικά προγράμματα ώστε κάθε χώρα να μπορεί να δημιουργήσει τις σχέσεις, του συνδέσμους μεταξύ πόλεων και ε, αγροτικών περιοχών, γειτονικών που έχουν μεν πόρου, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει δικτύωση. πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να διευκολύνουμε τη συνεργασία των ε, πόρων, των πόλεων με το ε, γειτονικό τους περιβάλλον. 5% λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε επίσης και το ITI. Απλά υπάρχει στεναρή αντίσταση από κάποια κράτη-μέλη εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον. Γι' αυτό προτείνουμε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ITI για αυτό το λόγο. Όχι όμως υποχρεωτικά. Και άλλες μέθοδοι μπορούν να βρεθούν. Και άλλου είδους ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση ε, ταμείων λέγαμε να ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα για 7 χρόνια στις πόλεις, αλλά υπήρξε η στεναρή αντίσταση από κάποιους. Γι' αυτό προτείνουμε να διαφοροποιήσουμε το επίπεδο ανάθεσης καθηκόντων για τις πόλεις ή για τις λεγόμενες αστικές λειτουργικές περιοχές. Για τις από απόκεντρες ε, περιοχές εκεί δεν έχω κάποια αλλαγή. Να προτείνω για να συνοψίσω στην πρότασή μου η γενική ιδέα είναι να παραμείνει θεματική συγκέντρωση, αλλά να καταστεί πιο ευέλικτη, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να επιλέξουν και να ορίσουν το περιεχόμενο, να διατηρήσουν με τη συγκέντρωση, αλλά να μην τα περιορίσουν όλα, να μην τα περιχαρακώσουν όλα, γιατί τότε περιορίζεται η ελευθερία και η ευελιξία. Και νομίζω ότι εν καιρό κρίσης θα πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό, ευέλικτο ε, και εύκολο να αλλάξει σύστημα. Και μιλάμε και για τον αναπρογραμματισμό που δεν είναι στο ε, Ταμείο Περιφέρειας Ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό για να μπορούμε να αναπρογραμματίζουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ, αυτά είχα να πω. Thank you, Ian, very much. Uh, Σας ευχαριστώ, Γιάν. Συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ φορτωμένη η ατζέντα μα σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα όλοι να με ακούσετε, να σεβαστείτε τον κανόνα ότι λέμε εξ αρχής ε, της συζήτησης ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Τώρα λοιπόν να δηλώσετε ποιος θέλει να πάρει το λόγο για την έκθεση του Γιάννη, γιατί στην περίπτωση αυτή θα μπορέσω να καταλάβω, ε, θα μπορέσω να αποφασίσω πόσο χρόνο θα δώσω τον καθένα σας. Τρεις εισηγητές όδης έχουμε. Δεν ξέρω, θέλει κανείς άλλος πέρα από τους κοιόδης να πάρει το λόγο, Κορνέλια τέταρτο άτομο. Κλείνω λοιπόν το κατάλογο των ομιλητών. Πέτερ Σίμον. Σάιμον. Νίλσεν, ο κύριος Νίλσεν. Ωραία. Κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών. Θα σας πω σε λίγο πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας, αλλά σκιώδη σας παρακαλώ να μην κάνετε γενικά σχόλια, να επικεντρωθούμε στις ε, λεπτομέρειες της τροπολογίας, τα επιμέρους στοιχεία. Η Κέρστιν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σωστά τα είπατε, είναι φορτωμένη η ημερήσια διάταξη, αλλά έγινε και η πρώτη συνάντηση των σκιωδών. Είναι η πρώτη περίσταση που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα γενικά. Θα είμαι αρκετά σύντομη. έχουν αναφερθεί τα σημαντικά στοιχεία για τους σοσιαλιστές. Χαίρομαι που ο εισηγητής σε αρκετά θέματα είναι κοντά στις δικές μας απόψεις. Να πω δύο λόγια για την υποστήριξη των υποδομών, όπου πάντα λέγαμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα και σε πιο πλούσιες περιοχές. Αυτό που σίγουρα ανέφερε και ο κύριος Όλμπριχτ είναι η υποστήριξη των μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί όντως οι προδιαγραφές είναι πάρα πολύ αυστηρές στην παρούσα φάση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει γενική απαγόρευση, γιατί χρειαζόμαστε τις ε, ενισχύσεις στους τομείς αυτούς, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλες είναι οι επιχειρήσεις, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχει διακριτική μεταχείριση και στη θεματική συγκέντρωση ε, είμαστε πολύ κοντά με τις απόψεις του κυρίου Ολμπρίχτ. Όντως, οι πιο πλούσιες περιφέρειες ε, θεωρούν ότι το 80% είναι πολύ ε, περιοριστικό στους θεματικούς στόχους επίσης θα πρέπει να ε, εργαστούμε προκειμένου στις προτεραιότητες ε, να ε, υπάρξει κάποια ισορροπία. Και βασική, βασικός όρος είναι οι ενισχύσεις των επιχειρήσεων. Και οι δημογραφικές αλλαγές και ο τουρισμός, ο πολιτισμός. Και θα ήθελα επίσης να επαναλάβω το εξής. Όσο σημαντική και αν είναι η επικέντρωση σε τρεις βασικούς στόχους, να μην ξεχνάμε και την κλασική, το κλασικό καθήκον των ταμείων αυτών που αναφέρονται και στο άρθρο 2. Η ιδέα του να συμπεριληφθούν οι αστικές συγκοινωνίες μικρής απόστασης στο στόχο 4 θεωρώ ότι είναι καλή και για την ενίσχυση των πόλεων, είναι σαφές ότι οι απόψεις μας συγκλίνουν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη σχετικών φόρουμ, αλλά και αξώνων προτεραιοτήτων. Όλα αυτά θα πρέπει να μείνουν σε επίπεδο δήμων, πόλεων. Ένα θέμα σε ό,τι αφορά την ε, προώθηση, την ενίσχυση κατασκευής αγωγών πετρελαίου. Εδώ δεν σύμφωνο. Στη θεματική επικέντρωση. Θεωρούμε ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στις περιφέρειες αν ένας τέταρτος στόχος πέρα από τους τρεις που ορίζονται θα μπορούσε να επιλεχθεί από κάθε περιφέρεια. Δηλαδή πέρα από τους τρεις υποχρεωτικούς στόχους να μπορεί κάθε περιφέρεια να επιλέγει και ένα τέταρτο στόχο δικό της. Ε, νομίζω ότι αυτό θα εγγυούταν την απαραίτητη ευελιξία. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε και θεωρούμε ότι θα είναι πολύ καλή, καλός ο κανονισμός. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαντέλη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για το σύνολο της εργασίας του και ε, για την καλή συνεργασία που είχαμε σαν ε, σκιώδης η πολιτιστική διάσταση μέσω των διαφόρων προτεραιοτήτων ε, επένδυσης είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και επίσης εξίσου θετικό ε, το ότι συμπεριέλαβε και την αστική ανάπτυξη καταδικάζοντας αυτή τη λεγόμενη πλατφόρμα υπάρχουν ε, οι οικολογικές δεσμεύσεις ε, και οι ε, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και ενεργειακές δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται και στην στρατηγική 2020. Γνωρίζουμε τα προβλήματα του ETS, των ποσοστώσεων εκπομπών και επίσης ε, αυτή η μείωση του κατά 20% της ε, κατανάλωσης ενέργειας χωρίς όμως να δούμε από πιο κοντά το θέμα της ενεργειακής ε, απόδοσης καθώς επίσης και η αύξηση της χρήσης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Το άρθρο 9 κατά την άποψή μου δεν έχει έννοια εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ποσοστά και για τις αυξημένα, για τις μεταβατικές περιοχές, καθώς επίσης και για τις πιο αναπτυγμένες περιοχές. Η μη δέσμευση σε αυτούς τους στόχους σημαίνει ότι σε τοπικό επίπεδο ε, θα στερήσουμε δεκάδες, εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Τέλος. Βλέπω ιδιαίτερα περίεργη αυτή την βούληση ε, να γίνουν δικαιούχοι, των, δηλαδή να, να η επιλεξιμότητα των ε, ταμείων σε πιο μεγάλες εταιρείες. Ενώ οι μικρές εταιρείες μέχρι τώρα τελικά ε, παίρνουν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των διορθωτικών ταμείων και ε, δεν έχουν αρκετούς πόρους αντίθετα από τις μεγάλες εταιρείες για να αναπτυχθούν παρότι παίζουν τόσο σημαντικό κινητήριο ρόλο. οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μικρές και οι μεσές, αν είχαν ιδιαίτερη και καλύτερη πρόσβαση στις, ε, στα διαφορετικά ταμεία τότε, και το έχω πει επανειλημμένα, τότε θα μπορούσαν πραγματικά να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το πραγματικό Small Business Act, δηλαδή ξεκινώντας από μικρός να ε, καταφέρεις να μεγαλώσεις και ε, νομίζω ότι η δικιά μας Επιτροπή μέσω του ΦΕΝΤΕΡ θα πρέπει να ενθαρρύνει αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά για τους ε, τρεις ομιλητές που έχουν μείνει. Κορνίλια. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, υπάρχει μία σειρά στοιχείων με τα οποία συμφωνούμε. Αυτό είναι σαφές και ως κοιόδης αποφασίσαμε και εμείς ε, οι υποδομές ε, θα πρέπει να επεκταθούν στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν θα πρέπει να εξαιρούνται, να αποκλείονται και θα πρέπει επίσης να κοιτάμε ένα κράτος μέλος και να περιφέρεια το τι υποστηρίζεται, τι ενισχύεται. Ε, συμφωνούμε για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό και τον τουρισμό για την ε, αστικέ κοινωνίε μικρή απόσταση, φυσικά και συμφωνούμε. Ενεργειακή αποδοτικότητα θα πρέπει να παραμείνει και θα πρέπει να το προσέξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πού είναι οι διαφορέ μας τώρα στους θεματικού στόχους. Ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου για όλα αυτά τα ποσοστά που αναφέρονται. Θεωρώ ότι όταν υπάρχουν θεματικοί στόχοι θα πρέπει να αξιοποιούνται. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γιατί κάποιο θεματικό στόχος θα πρέπει να λαμβάνει κάτι λιγότερο στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 όλοι εκεί δεν εντάσσονται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει γενικά και να γίνει ένα σημαντικό βήμα για την αστική ανάπτυξη, για την προσέγγιση που υποστηρίζεται την, ε, μας βρίσκει σύμφωνους. Ε, τα συζητήσαμε και εκτενώς ε, στα προηγούμενα, στις προηγούμενες συνεδριάσεις για τους αγωγούς τους πετρελαϊκούς και για τον καπνό. Δεν συμφωνούμε, λυπάμαι, αλλά νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουμε να συμφωνήσουμε. Θα δούμε και τις τροπολογίες. Ελπίζω να χαρείτε με τις τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο κύριος Σάιμον. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συνεδρίαση και την παρουσίαση για τις λειτουργικές ε, αστικές περιοχές για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη που δεν σταματάει στα όρια των πόλεων που μπορεί να περιλάβει και διάφορες, ε, διάφορους δήμους σύμφωνο Και κάνω και ένα βήμα παραπάνω για να λαμβάνουμε υπόψη πιο πολύ τα διάφορα μοντέλα αστικής ανάπτυξης και να δώσουμε και πιο πολύ ευελιξία σε αυτό το νέο μέσο, θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε τους λειτουργικούς αστικούς χώρους και να τους επεκτείνουμε με άλλους ε, λειτουργικούς χώρους, λειτουργικές περιφερειές. Για παράδειγμα, ε, στην περίπτωση του τουρισμού υπάρχουν ε, διάφοροι χώροι, διάφορες περιφέρειες οι οποίοι έχουν τη σημασία τους στην, ε, στον τουρισμό. Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επέκταση και θα υποβάλω σχετική τροπολογία και ελπίζω μέσω συζήτηση να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε. Μια άλλη παρατήρηση σε ό,τι αφορά το 5% για τις ενοποιημένες περιφερειακές επενδύσεις. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μήπως και αυτό δεν θα έπρεπε να ορίζεται σε επίπεδο εθνικού κράτους μέλους, αλλά σε επίπεδο λειτουργικού προγράμματος και παράλληλα να σκεφτούμε μήπως οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι οποίοι έχουν την αναλογή δομή και πρόθεση και θέληση, μήπως θα μπορούσαν να αναλάβουν τη διαχείριση των ITs, προκειμένου και αυτή η μέση διαχείριση να είναι ευθύνη τους. Και νομίζω ότι και αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλσον για δύο λεπτά. Θα είμαι πάρα πολύ συντομός να στηρίξω τον εισηγητή και έχοντας ε, την ε, εμπειρία ε, των αδειοκατοικημένων βορείων περιοχών ε, τον ευχαριστώ γιατί ε, έχει βάλει στην έκθεση και τη διάσταση του πολιτισμού και του αθλητισμού ε, γιατί σε μερικές περιοχές αυτή είναι η μόνη δυνατότητα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το δεύτερο σημείο είναι οι υποδομές. Είναι δύσκολη η συζήτηση για τα θέματα αυτά γιατί εμπλέκονται πάρα πολλά χρήματα εξορισμού πάντως ε, μπορεί οι βόρειες περιοχές, οι δικές μας, να είναι παραδοσιακά ε, πλούσιες, όμως είναι τόσο αραιοκατοικημένες ε, που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Η ευρυζωνικότητα λοιπόν είναι ένα σημαντικό θέμα και τέτοιου είδους υποδομές θα πρέπει να στηρίζονται. Επίσης μπορεί να γίνει και κάποια στρατηγικά στοχευμένη δουλειά για τον τουρισμό. Ευχαριστώ λοιπόν για τα δύο αυτά σημεία. Νίκολας Μάρτιν από την Κομισιόν. Τρία λεπτάκια το πολύ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι κάποια από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει στην έκθεσή του εισηγητή ε, ήδη αναφέρονται στην έκθεση επιτροπή, ε, κυρίω όσον αφορά ε, την αστική διάσταση. Εκεί διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για διεύρυνση των δυνατοτήτων. Εμεί θα προτιμούσαμε απλή αναφορά σε urban areas και όχι functional urban areas, γιατί υπάρχει και η, ακόμα ενδυνατότητα κοινά δυνατότητα χρήσης ε, της ε, πλατφόρμας οι περιοχές ε, οι οποίες όντως παρουσιάζουν προβλήματα σε σχέση με την ε, πρώτη επιτροπή, Επιτροπής ε, ε, σχετίζονται πρώτον με τη διεύρυνση του, του πεδίου εφαρμογής. Η διεύρυνση λοιπόν σε μεγάλες επιχειρήσεις αντιτίθενται στην ιδέα την οποία έχει η Κομισιόν όσον αφορά την δυνατότητα στήριξης, στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, και επίσης ε, μέσω της ε, διεύρυνσης της R&D. Στην προκείμενη όμως τροποποίηση προτείνεται απλά η διεύρυνση χωρίς εξειδίκευση. Επίσης, οι πιο αναπτυγμένες περιοχές, ε, λέει η εμπειρία μας, έχουν ήδη ε, κάποια ε, υποδομή, παρόλα αυτά δίνει, έχει περιθώριο για μια επιπλέον ανάπτυξη της υποδομής σε αυτές τις χώρες και τις περιοχές. Όσον αφορά τώρα τον καπνό και τον αποκλεισμό, Απλώς θέλαμε να δείξουμε ότι δεν θα υπάρξουν επενδύσεις στην καπνοβιομηχανία και αυτή είναι μια εναρμονισμένη ε, ε, ενωσιακή προσέγγιση. Όσον αφορά τώρα τον αθλητισμό και το, την κουλτούρα και τον πολιτισμό, αυτά τα στοιχεία δεν χρειάζεται κατά την άποψη της Επιτροπής να αναφέρονται. Ε, η Επιτροπή θεωρεί ότι εν γενός οι περιφέρειες μπορούν να αναπτύξουν τέτοιες δραστηριότητες. Πρόκειται για περιοχές επενδύσεων που βεβαίως μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία όσον αφορά ε, την ε, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, αλλά δεν υπάρχει λόγος στα στοιχεία αυτά να υπάρξει ε, αυξημένη παρέμβαση Ευρωπαϊκής, σε, της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το ETS. Θεωρούμε ότι μεγάλες διευρύνσεις μπορεί να δυναμητήσουν το σύστημα ETS. Και δύο ελάσσονο σημασία στοιχεία όσον αφορά την θεματική συγκέντρωση. Εδώ η εισηγητής ε, ε, θέλει τρία πράγματα να μειώσει τα ποσοστά να αυξήσει ε, την, ε, τις, ε, τα θεματικά ποσοστά τα οποία μετρούν καθώς επίσης να λάβει υπόψη και την αστική κινητικότητα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι με τέτοια διήθηση και διάχυση το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Επίσης, η διατύπωση των ε, προτεραιοτήτων ε, επενδύσεων. Μην ξεχνούμε ότι οι θεματικοί στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν ε, τις επενδύσεις. Μπορούν να αποσαφινιστούν, αλλά δεν θα πρέπει να διευρυνθούν, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε την εστίαση την οποία αποζητούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Νίκολας. Γιάννη, δύο-τρία λεπτά έχεις για να απαντήσεις. Δηλαδή καλύτερα είναι να επικεντρωθεί σε, αυτό, αυτά με τα οποία συμφωνείς από αυτά που άκουσες. Στις κοινωνικές επιστήμες η διορθωτική φιλοσοφία σημαίνει ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στην πολύ βαθιά δομή. Στη βαθιά δομή λοιπόν ε, συμφωνώ με πολλούς ε, με τους οποίους ενδεχομένως στην επιφάνεια δεν θα συμφωνήσω. Εν πάση περιπτώσει. Γενικώ, να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στη συζήτηση για τις επικοδομητικές παρατηρήσεις οι οποίες καταδεικνύουν και τις διαφορές που έχουμε ας πούμε με την Κομισιόν γιατί η πρώτη αντίδραση των συναδέλφων ε, ήταν ότι θα πρέπει ε, αυτού του είδους οι επενδύσεις να ε, ειδωθούν ε, σαν μέρος της οικονομίας και των επενδυτικών διεργασιών και όχι σαν αλλαγή της ζωής. In ε, και ούτε ή άλλως εδώ δεν είναι η ολοκλήρωση και το επιστέγασμα, είναι η αρχή των διαπραγματεύσεων. Θα έχουμε και τις επαφές με τα κράτη-μέλη. Ε, είναι εκπληκτικό το ότι τα κράτη-μέλη τα οποία ε, δεν συμφωνούν με την συνοχή, είναι anti-cohesion, είναι, αυτά τα οποία είναι αυτά τα οποία συμφωνούν με την προσέγγιση μου. Και δύο παρατηρήσεις, κυρία Πρόεδρε, πιο γενικού χαρακτήρα. Η γενική στάση, η φύση της έκθεσής μου είναι ότι πρέπει να αποφασίζουμε ε, δεν πρέπει να αποφασίζουμε για τις λεπτομέρειες της Βρυξέλλες, δηλαδή να καταρτίζουμε κάποιους γενικούς στόχους, κάποιες γενικές γραμμές και μετά ε, οι περιοχές, οι περιφέρειες να βρίσκουν μόνες τους πώς μπορούν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται, θέλουν να επιτύχουν τους τρόχους αυτούς. Γιατί εάν περιγράψουμε σαφέστατα τα πάντα, το περιθώριο ελιγμού είναι πάρα πολύ μικρό. Θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Ε, αλλά αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ονομάζει διήθηση ή διάχυση. Δεν, δεν έχουμε λοιπόν την ίδια άποψη. Ας είμαστε επομένως πιο αυστηροί. Ας είμαστε πιο ε, αυστηροί όσον αφορά την ερεσιμότητα, όσον αφορά τα κριτήρια, όσον αφορά την, ε, τους ελέγχους. Ε, αλλά να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί θέλουμε ας πούμε περισσότερες δουλειές, ας δούμε τότε ποιος μπορεί να δημιουργήσει τις περισσότερες θέσεις εργασίας αλλά σε μια χώρα μπορεί να υπάρχει μια επιχείρηση η οποία να έχει δημιουργήσει ήδη ε, πολλές θέσεις εργασίας και να μην είναι και μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά να βοηθάει την περιφέρεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι δύο λέξεις, ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Το πώς θα το επιτύχουμε αυτό, αυτό είναι το σημαντικό. στην ουσία δεν διαφοροποιείται πάρα πολύ η άποψή μας. Διαφοροποιείται η αντιμετώπιση της μεθοδολογίας μέσω της οποίας μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι. Θα συνεχίσουμε να βεβαίως να συζητούμε το θέμα και το πρόβλημα του ETS. Ε, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται ότι τις λεπτομέρειες του ETS. Ε, δεν θέλω να συζητήσω το θέμα του καπνού. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι στο EDRF. Από τη στιγμή που αναφέρονται γενικά στοιχεία της ε, ενωσιακής ε, πολιτικής. Λέμε ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις, ιδίως δε μέσω του ERDF. Γιατί, δεν το καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ως αρχή είναι καλή η θέση μας, γιατί αν έχουμε πλήρη συμφωνία εξ αρχής, τι θα διαπραγματευτούμε. Επομένως θεωρώ ότι τώρα είμαστε σε μια καλή θέση. Ε, κάποιες χώρες μέλη και οι Κομισιόν βεβαίως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια σημεία της θέσης τους. Και να προχωρήσουμε λοιπόν. Ε, α, οι υποδομές επίσης. Ε, ακόμα και σε αναπτυγμένες περιοχές ένα κομμάτι της υποδομής μπορεί να είναι απολύτως καινοτόμα και να δημιουργήσει νέα στοιχεία ε, και θα δώσει τη δυνατότητα και, μάλλον γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν. Δεν μπορεί να κλείσουμε τις πόρτες από την αρχή. Η γενική φιλοσοφία λοιπόν είναι ε, να γίνουμε πιο ανοιχτοί, πιο ευέλικτοι και μετά να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που είναι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι θα ήθελα να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό, αν και φαντάζομαι ότι θα τεθούν και κάποια γενικά θέματα στις επερχόμενες συζητήσεις, επειδή ε, δεν έχει έρθει ακόμα ο κύριος Τσέλερ για την επόμενη έκθεση θα ήθελα να ξεκινήσουν οι συγητές για το γενικό κανονισμό. Η εστίαση σήμερα θα είναι στο στρατηγικό πλαίσιο, αν και φαντάζομαι ότι θα θέλετε να παρουσιάσετε και τις τροπολογίες οι οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμα στην, στο σχέδιο έκθεσης. Ό,τι πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να κάνετε για το θέμα αυτό. Για το 12 λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον ε, Λάμπερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρο και συγχαρητήρια που καταφέρατε στην πρώτη ώρα να φτάσετε στο σημείο 12. Ναι, μπορεί να πάω και πιο γρήγορα, αν θέλετε, λέει η Πρόεδρο, σω να ε, ακολουθείτε το πνεύμα των τελευταίων ημερών, για να σοβαρευτούμε. Ναι, είμαστε σε φάση εξέταση και έχουν γίνει συζητήσει βήμα προ βήμα για το σχέδιο το έγγραφο εργασίας, μπορούμε να συζητήσουμε για το πρώτο, αν θέλετε, για τις πρώτες τροπολογίες και χαίρομαι που τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμα και στο Στρασβούργο, καταφέραμε να συζητήσουμε με τους ε, εισηγητές ε, που, μας, ε, που κατάφεραν να έρθουν τις τροπολογίες γιατί αυτό κατέδειξε ότι αν κάτσουμε και συνοηθούμε και τον προτέρων, μπορεί τελικά να μην ε, υποβληθούν 2.000 τροπολογίε. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο φυσικά. Αν λοιπόν ακολουθούμε τη διαδικασία που ακολουθήσαμε, βήμα προς βήμα, προσπαθούμε να συνοηθούμε εξ αρχής, προκειμένου να γίνει ψηφοφορία αρχές Ιουλίου, αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί, γιατί όπως είπε ο Γιάννα Όλμπριχτ, δημιουργείται έτσι ένα πλαίσιο για τη συζήτηση, προκειμένου να συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο στη συζήτηση. Γιατί μόνο με την ψηφοφορία για τον κανονισμό μπορούμε να τοποθετηθούμε, αν θέλετε, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί υπάρχει και μία τάση στο Συμβούλιο, ξέρετε, θα το συζητήσουμε και πιο μετά με τον Επίτροπο και με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας για την πρότασή τους και την πρόοδο που σημειώνουν. Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα έχουν αποφασιστεί ομόφωνα κάποια ζητήματα στο Συμβούλιο και θα μας πούν ότι Α, δεν μπορούμε εκ των, εκ των υστέρων να τα ξανανοίξουμε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συναπόφαση. Άρα σας παρακαλώ συνάδελφοι, προσέξτε, διαβάστε τις τροπολογίες μας, προτού καταθέσετε νέες τροπολογίες. Μην υπάρχουν ε, διπλές ε, τροπολογίες και επικαλύψεις. Να προσέξετε παρακαλώ. Εντάξει, μην ε, φοβηθείτε κιόλα, αλλά μην καταθέτουν όλοι ολόκληρες ε, σειρές τροπολογιών. Και κάτι άλλο. Πρόεδρε, ναι. Σήμερα, σύμφωνοι μαζί με την Κωνσταντσε, ας προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στο CSF, που έχει μια δική του πλέον διαδικασία και μπράβο μας, γιατί το πολεμήσαμε προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο διατυπώνεται ήδη σε άρθρα και μπορεί να, τροπο, να τροποποιηθεί. Και αυτό καταδεικνύει γιατί αγωνιούσαμε να μπει στο νομικό κείμενο. Γιατί μας διευκρινίζει πώς λειτουργούν όλα αυτά τα άρθρα στην πράξη και πώς θα πρέπει να γίνουν κατανοητά. Αυτό είναι σημαντικό για να καταστεί απτή η πολιτική μας και για να καταστεί και επικοινωνιακή η πολιτική μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τις εποχές αυτές που μιλάμε για την ανάπτυξη, για την ε, δημιουργία θέσεων εργασίας. Πολλά τροποποιήθηκαν στις διαδικασίες για να υπάρχει πιο μεγάλη συνεργία παραποτέ. Αλλά καταλαβαίνω ότι αν ε, παρουσιαστεί το CSF ως τροπολογία, θα πρέπει να υπάρχει και λίγο πιο πολύ χρόνος για να το εξετάσουμε. Εμείς αποφασίσαμε να δώσουμε μία εβδομάδα παραπάνω. Είναι μία τροπολογία την οποία μπορείτε να διαβάσετε και ευχαρίστως να σας την διευκρινίσουμε, να σας την εξηγήσουμε και στους κοιότης, αλλά και σε οποιονδήποτε το επιθυμεί. για όποιον θέλει. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν σήμερα. Και να πω και δύο λόγια, κοιτώντας και προς την πλευρά της Κωνσταντσε. Φυσικά και στα κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο. Το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε τα οριζόντια ζητήματα και τις εγκάρσεις προκλήσεις. Το θέμα είναι οι συνέργειες, η συντονισμός των ε, ε, κονδυλίων σε ό,τι αφορά τους στόχους του 2020. Όλα αυτά είναι πολύ απαραίτητα. Το θέμα λοιπόν είναι το CEF, οι σημαντικές υποδομές, τα σημαντικά έργα υποδομών, τα νέα μέσα NP, NPDF, εκτός συνόρων. Το θέμα λοιπόν είναι το πώς θα εφαρμοστεί ακριβώς αυτός ο συντονισμός. Άρα, για να μην επαναλάβω θέματα περιεχομένου, θα ήθελα απλά να τονίσω ποιος είναι ο απότερος στόχος της δουλειάς μας των τελευταίων εβδομάδων. Και εδώ θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής. Κωνσταντζε, εξετάσαμε και κάποιες εις βάθος τροπολογίες, όχι για να προσθέσουμε νέα στοιχεία, αλλά για να διευκρινίσουμε νομικά ζητήματα τα οποία ε, έπρεπε να διευκρινιστούν από τις νομικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και θα, κατα... θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες για να διευκρινιστούν περαιτέρω κάποια θέματα. Αυτό θα ληφθεί υπόψη και αργότερα στη μετέπειτα φάση Εξέταση των τροπολογιών. Oh, this is the information. Constanza, can you help me out? Κωνσταντσα, τι έχει να μας πει. Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Η Πρόεδρος επιτρέπει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να συμπληρώσω. Ίσως το θέμα των τροπολογιών, τις οποίες ανέφερε ο Λάμπερτ προς το τέλος, νομίζω ότι ένα πολιτικό σημαντικό θέμα για μας είναι η εισαγωγή του κώδικα δεντολογίας, του κώδικα συμπεριφοράς. Αυτό ως κοινοβούλιο μας απασχολεί ιδιαίτερα, θα πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί θα πρέπει να καταδείξουμε ότι θέλουμε να υπάρξει κώδικας δεοντολογίας, ε, ότι θα πρέπει να διευκρινίζεται και η καλή διακυβέρνηση και η αρχή εταιρική σχέσης. Υπάρχουν και τεχνικές τροπολογίες, οι οποίες όμως είναι σημαντικές ε, για το Common Strategic Frame, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Οι συνάδελφοι από τη Γραμματεία πραγματικά έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Να σας ευχαριστήσω όλους όσοι καθίσατε και βλέπατε επί ώρες, γιατί τα κείμενα τα οποία είχαμε προτείνει τελικά ε, τα επεξεργαστήκατε με τέτοιο τρόπο. Λάβατε και ένα email για το πώς θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές. Νομίζω ότι αύριο θα λάβετε και ένα email όταν μας διευκρινίσει η νομική υπηρεσία ποια θα, θα πρέπει να είναι η ακριβής διατύπωση για το Common Strategic Frame. Ένα σημαντικό σημείο πήραμε, το πρώην κεφάλαιο 4, γιατί είπαμε ότι στην παρούσα φάση δεν βλέπουμε ότι υπάρχει επιπρόσθετο όφελος να υπάρξει συντονισμός των θεματικών στόχων ανά άξονες προτεραιοτήτων, αλλά νομίζω ότι τα υπόλοιπα τέσσερα καλό είναι να μείνουν στο κόμμα στο strategic frame όσο έχουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Στο θέμα τώρα του τι θα κάνουμε με τις τροπολογίες να σας παρακαλέσω όντως, ε, πέρα από αυτά που είπε ο Λάμπερτ, να σας παρακαλέσω το εξής. Στη παρούσα φάση, πολλοί ψάχνουν ε, ε, βουλευτές από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για να τους μιλήσουν και θα είχε νόημα αν οι συνάδελφοι υιοθετήσουν τροπολογίες του Συμβουλίου και τις καταθέσουν, αλλά αυτό θα μας αφαιρούσε, αν θέλετε, διαπραγματευτική ικανότητα. Γιατί οι διαπραγματεύσεις τα ψέματα πώς κινούνται, κάτι σου δίνω εγώ, κάτι μου δίνεις εσύ. Αν εξ αρχής έχουμε υιοθετήσει κάποιες απόψεις τους, δεν έχουμε διαπραγματευτικό περιθώριο, δεν μπορώ να σας το πω πιο καθαρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, Ξέρετε ότι χρειαζόμαστε αυτό το διαπραγματευτικό περιθώριο και όπως είπε και ο Λάμπερτ, όπως είπε και ο Γιάννα άλλωστε, βρισκόμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων στις 9 Ιουλίου όταν θα ψηφίσουμε. Άρα αυτή την ιστορική ευκαιρία που μας δίνεται για την περιφερειακή πολιτική στα πλαίσια της συναπόφασης θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε και θα πρέπει να πω και το εξής για το Common Strategic Frame είναι πραγματικά νέο έδαφος. Για πρώτη φορά ε, κάνουμε και λαμβάνουμε ίδια πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο και προτείνουμε νέα νομοθεσία. Αυτό είναι κάτι καινούργιο, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Να δούμε πώς θα ψηφιστεί και να φροντίσουμε να είναι σωστή και καλή η διαπραγμάτευση κυρίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντσε. Δύο ε, δύο σκέδες συζήτηση έχουμε. Ευχαριστώ. Πραγματικά πολύ καλή συζήτηση είχαμε στο Στρασβούργο. Εκεί διευκρινίστηκαν πολλά θέματα. Και τέθηκαν και πολλά ζητήματα επιτάπτους του συναδέλφους. Πολλές φορές είναι ενδιαφέρον να ξέρουμε και τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Θα ήταν ενδιαφέρον λοιπόν αν κάποιος έχει κάποια διασύνδεση με κάποιο υπουργείο, με τις κυβερνήσεις, διότι πλέον ολοκληρώνεται, αν θέλει, και το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, το κουτί, το διαπραγματευτικό. Και αν κάποιος ε, έχει κάποιες πληροφορίες, είναι νομίζω πολύ ενδιαφέρον. Ε, παραδείγματος χάρη έχουμε το παράρτημα 2, μας έστειλε μια λευκή σελίδα η Κομισιόν, αλλά η Προεδρία και τα κράτη-μέλη κυρίως με αυτό ασχολούνται. Δεν ξέρω αν κάποιοι γνωρίζουν περισσότερα από εμένα. Υπάρχουν θέματα λοιπόν που δεν τα γνωρίζουμε και τα οποία είναι διαπραγμάτευση. Πάντως αυτό που συζητάμε κυρίως ε, δεν έχει φύγει. Δεν ξέρω μήπως υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Ίσως ήταν καλό να τα προσθέσουμε από τη μία βλέπουμε να συζητείτε το χρηματοοικονομικό σκέλος ε, και εμείς συζητούμε το θεματικό σκέλος. Καλό θα ήταν να συζητήσουμε αυτά ταυτόχρονα. Παραλαμβάνω όμως ότι υπάρχουν κάποια κενά. Αυτό που θέλω εγώ να τονίσω. Ε, δεν έχω κάποια στοιχεία για την 1η Μαΐου, για το, τον πίνακα αυτόν. Αλλά υπάρχουν σημαντικά ποσά. Δεν ξέρω αν έχει ανοίξει προθεσμία για τα διάφορα ταμεία, το κοινωνικό ταμείο κτλ. Είναι και ένα άλλο θέμα που δεν έχουμε συζητήσει, ακόμη θα συζητηθεί όμως ε, στην Επιτροπή Προαπολογισμών, το υπόλοιπο προς εκαθάριση. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό για να ολοκληρώσουμε τις προοπτικές του 2013 και επηρεάζει πάρα πολύ και το νέο πολιτές ε, πλαίσιο, δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το τεράστια ποσά, 200-209 δις ευρώ. Αυτό το υπόλοιπο προς εκαθάριση είναι πολύ σημαντικό. Κάποιοι λένε δεν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά αν δούμε τον κανονισμό 1083 υπάρχει προθεσμία νήσιν 2 νήσιν 3. Κάποιες χώρες μπόρεσαν πέρυσι να εκπληρώσουν το νήσιν 2. Έχουμε οικονομική στενότητα, ε, πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Εγώ συμφωνώ με αυτό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, το CSF. Το διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά, είναι στο παράρτημα και σωστά. Δεν έχει την ίδια νομική ισχύ με το βασικό κανονισμό. Στηρίζω λοιπόν το γεγονός ότι βρίσκεται σε παράρτημα, αλλά να τίθεται εγώ όμως είμαι υπέρ. Και το δεύτερο που θέλω να αναφέρω είναι δεν ξέρω ποια θα είναι η εκβασή. Αυτή τη έκθεση Communication Europe. Θα δούμε τι ακριβώς θα προκύψει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Θα κάνουμε τις προσπάθειες μας, νομίζω όμως ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Έτσι έχουν τα πράγματα βέβαια. Πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο το πώς ε, και το πού θα πηγαίνουν τα χρήματα. Ξέρουμε ότι το 10% θα μπει σε έναν πίνακα. Και αν κάποιος είναι καλός μπορεί να έχει πρόσβαση, κάποιος άλλος όχι. Δεν θα μπει δηλαδή στον Ταμείο Συνεχής και θα είναι τόσο απλά τα πράγματα. Συμφωνώ και με την Κωνσταντσε ότι υπάρχει και πολύ μεγάλη άσκηση πίεσης από λόμπι. Αλλά earmarking, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν υπάρχει. Καλό θα ήταν να μπορούσαν αυτά τα έργα να καλύψουν 27 κράτη-μέλη, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επαρκούν τα χρήματα για αυτό το σκοπό. Το τελευταίο πράγμα που συζητήσαμε, η πρόταση της Κομισιόν για το ΦΠΑ. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα, Έχουμε την φυστάμενη κατάσταση και έχουμε και την ε, πρόταση των συγητών. Τρεις είναι οι δυνατότητες. Είτε να μείνουν τα πράγματα ως έχουν, είτε το άρθρο 55 παράγραφος 3c ε, την πρόταση Κομισιόν να ε, την εγκρίνουμε ή τρίτη επιλογή να στηρίξουμε τους εισηγητές μας. Εγώ τίνω να ε, ταχθώ υπέρ της θέσης των εισηγητών γιατί θα έχουν πιο πολλούς πόρους έτσι οι δικαιούχοι και έτσι θα μπορούν να υλοποιηθούν τα ταμεία, συνοχή τα διορθωτικά ταμεία. Βέβαια είναι πολύ πλοκό το ζήτημα. Είναι σημαντικό το ζήτημα. Θα ήθελα να υποστηρίξω λοιπόν εδώ τους εισηγητές. Σας ευχαριστώ. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριος Βλάσακ. Αν με επιτρέπετε, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε ορισμένε από τις ε, πτυχές που πρέπει κάπως να οριστικοποιηθούν. Πρώτα απ' όλα. Αυτό το performance reserve δεν δίνει επαρκή κίνητρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο αυτό παθηματικό και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, με τρόπο αποτελεσματικό. Τώρα στο ΦΠΑ ε, έκαναν και άλλοι συναδελφοί σχετική αναφορά. Η επιλεξιμότητα κτλ. Όλα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατά την άποψή μου στο πολιτές πλαίσιο. Στο γενικό κανονισμό και να υπάρχει ένας κανόνας νη χ, εν x. Τώρα, πώς αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται. Δεν θα πρέπει να είναι τόσο αυστηρός ο προσδιορισμός. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερη ευελιξία. Σε εθνικό επίπεδο. Τώρα το ανώτατο όριο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Δύο είναι οι επιλογές. είτε να καθοριστεί ένα ενιαίο επίπεδο για όλα τα είδη περιφερειών, είτε να αυξηθούν τα, περιφέρ τα ποσοστά για κάποια είδη, κάποια τύπους περιφερειών. Ίσως αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των συμφωνίων εταιρικής σχέσης. Σε όλους τους στόχους, πιστεύω, για όλα τα ταμεία, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση του ανώτατου ποσοστού συγχρηματοδότηση, 85%. Τελευταίο σχόλιο. Σχέση μεταξύ τα συνοχής και άλλων προγραμμάτων όπως ορίζον 2020. Θα πρέπει να είναι εναρμονισμένα αυτά. Κατά τα άλλα συμφωνώ με τη συζήτηση. Πρόεδρος, κλείνω εδώ το κατάλογο των ομιλητών, αγαπητοί συνάδελφοι η Κορνέλια και μετά ο Πέτερ. Δύο λεπτά σας παρακαλώ. Να ξεκινήσω α, με αυτό που μας απασχολεί πιο πολύ, όπου δεν ξέρουμε και πώς ε, να συμπεριφερθούμε. Η ρεσιμότητα εξάντε με απασχολεί ιδιαίτερα. Είτε να διαγραφούν όλα είτε να παρέμβουμε δυναμικά. Τι να σας πω, εμένα δεν με ικανοποιεί καθόλου, σας το λέω ξεκάθαρα. Και δεν βλέπω αυτή τη μεγάλη προστιθέμενη αξία πού βρίσκεται αυτό το επιπλέον όφελος και επί τις, αρχές έχουμε, τις αρχές έχουμε πρόβλημα με το σύστημα κυρώσεων. Και μάλιστα όταν δεν έχει σχέση με την ε, πολιτική συνοχή και σε ό,τι αφορά εξάντε περιπτώσεις ε, να το σκεφτούμε λοιπόν αυτό για τους γνωστούς λόγους. Για τον κώδικα απεντολογίας. Ναι, πολύ σημαντικός. Σκεφτήκαμε κατά πόσον θα έπρεπε να υπάρχουν πράξεις καταξιοδότηση. Αποφασίσαμε να... ότι μπορούμε να το αποτεχτούμε. Αλλά να ακούσω και άλλες απόψεις αν υπάρχουν. Υποστηρίζουμε τον εισηγητή για το στρατηγικό πλαίσιο, για το GSR και θεωρώ ότι είναι καλές ε, οι αρχές που περιλαμβάνονται και σας συγχαίρω. Είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με θέματα πιστοποίησης ε, και κλεισίματος των λογαριασμών. Πάρα πολλοί μας το έχουν πει ότι στο κλείσιμο των λογαριασμών ε, με μια καταληκτική ημερομηνία το πρόβλημα είναι ότι μετά από την ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να γίνει απολύτω τίποτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Του δυσκολεύει πάρα πολύ και τι προώθει τελικά να γίνεται project για ένα μόνο έτο. Αυτό δεν μπορεί να αποτελεί τον απότερο στόχο μας. Λοιπόν, κάτι θα πρέπει να κάνουμε στο πλαίσιο αυτό. Σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν ξέρω αν τα έχουμε συζητήσει όλα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί καλό είναι ότι υπάρχουν νέα χρηματοοικονομικά μέσα, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι που ενέχονται. Αυτά. Thank you, Peter Simon. Ο κύριο ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο πτυχές θέλω να τονίσω. Όπως αναφέρθηκε, καλώς ορίζω την ε, υποστήριξη διαχείρισης σε πολλαπλά επίπεδα για να τονιστεί και η σημασία και της τοπικής και της περιφερειακής ε, διάστασης σε όλες τις φάσεις. Τώρα σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της αρχής αυτής θα ήθελα να μιλήσω ότι δεν μπορεί ο κώδικας να αναπτυχθεί μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια ελάχιστα κριτήρια για την εταιρική σχέση, τα οποία θα πρέπει να μπουν και να ληφθούν υπόψη στα προγράμματα. Και κατά δεύτερον, θα ήθελα να μιλήσω για την απλοποίηση των κανόνων. Ε, επειδή το θέμα αυτό στην Επιτροπή το έχουμε συζητήσει σε πολλές περιπτώσεις και έχουν έρθει και πολλοί εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή μας, κοιτώντας τις προτάσεις που έχουν γίνει. είναι λίγο ύποπτο ότι δεν πρόκειται για απλοποίηση, αλλά ουσιαστικά μπορεί το αποτέλεσμα είναι προστιθέμενη γραφειοκρατία με τις προτάσεις αυτές ε, των εισηγητών σε ό,τι αφορά την υποχρέωση ελέγχου, την υποχρέωση αναφοράς. Θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα έρθει σύντομα επίτροπος Χαν και θα κάνει και σχετικές παρατηρήσεις, φαντάζομαι και επ' αυτού ε, στην επιτροπή σας, δηλαδή επί του CSF, του κοινού στρατηγικού πλαισίου και δεν θα ήθελα να προκαταλάβω ή να προδικάσω αυτά που θα πει ο ίδιος. Βέβαια, είδαμε το σχέδιο εγγράφου το παράρτημα είναι πρόσφατο σχετικά και δεν είχαμε την ε, δυνατότητα να το εξετάσουμε αναλυτικά και λεπτομεριακά. Θα ήθελα να περιοριστώ λοιπόν ε, σε λίγα σχόλια σε σχέση με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα, το έγγραφο έχει σχέση με προτάσεις τροποποίησης ε, και σε σχέση με τον ορισμό του CSF, του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Μία παρατήρηση λοιπόν θέλω να κάνω ενδέχεται να υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις για το ρόλο αυτού του πλαισίου. Συντονισμός και εξισορρόπηση των προτεραιοτήτων επενδύσεων. Αυτό λέει τροποποίηση, η τροπολογία. Και φαίνεται ότι έχει σχέση και με τη διαγραφή των βασικών δράσεων key actions που περιλαμβάνει το έγγραφο της Κομισιόν. Σίγουρα πρόκειται για ε, στόχους συγκεκριμένους ε, ε, για το Ταμείο Συνοχής, αλλά ε, σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, εδώ βλέπω θα καλυφθούν και τα πέντε ταμεία. Δεν γίνεται αυτό. Δεύτερον, υπάρχουν θεματικοί στόχοι, είναι ένα υποσύνολο, αν θέλετε, αυτών των στόχων, αυτές τις προτεραιότητες επενδύσεων. Εμείς από πλευράς ε, Κομισιόν θεωρούμε ότι ένας από τους πρωταρχικούς ρόλους ε, του πλαισίου, του στρατηγικού πλαισίου είναι να δίνει κάποια καθοδήγηση για το πώς τα πέντε ταμεία μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων αυτών ε, στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Και σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ορίσει αυτές τις, τις κύριες δράσεις, key actions, συγκεκριμενοποιώντας δηλαδή πώς τα πέντε ταμεία μπορούν να στηρίζουν διαφορετικού είδους επενδύσεις ε, ε, χωρίς ένα κοινό στόχο. Τώρα, αν μου επιτρέπετε να αναφέρω κάτι σε σχέση με τις ε, τροπολογίες για τον ίδιο τον κανονισμό των κοινών διατάξεων. Δεν έχει αναφερθεί από τους ε, συναδέλφους σας, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη διαγραφή του άρθρου 20 σε σχέση με το λεγόμενο performance framework, το πλαίσιο επιδόσεων βλέπουμε ότι ζητείται διαγραφή και του άρθρου 18 για το αποθεματικό και του άρθρου 20 για το πλαίσιο. Και υπάρχει κάποια διασύνδεση των δύο. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στους συζητητές σας να εξετάσουν πολύ καλά αυτό το θέμα. Εμείς μιλάμε για το performance framework. Το πλαίσιο είναι το σημείο αφετηρίας για μας. Είναι βασικό στοιχείο για την επίτευξη των αποτελεσμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αποθεματικό, το Performance Reserve είναι ένα από τα στοιχεία που είναι απόρρια τη εφαρμογή του πλαισίου. Δίνει κίνητρα για να υπάρχουν καλέ επιδόσει, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με αυτό το πλαίσιο επιδόσεων. Παραδείγματο χάρη, υποσκεκριμένε συνθήκε, αναστολή πληρωμών ή διόρθωση ε, στο κλείσιμο του λογαριασμού. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό το πλαίσιο. Το πλαίσιο επιδόσεων, όχι το αποθεματικό. είναι μοχλός για την εφαρμογή, τη διάρθρωση των προγραμμάτων και την επικέντρωση στα αποτελέσματα. Νομίζω θα ήταν απώλεια η διαγραφή του πλαισίου αυτού. Θα ήταν ουσιαστικά υπονόμευση ενός βασικού ε, σημείου. Θέλουν οι συγητές, λέει η πρόεδρος, να δευτερολογήσουν. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ίσως το βασικό σημείο είναι ότι η διαδικασία πλέον στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι. Θέλουμε να υπάρχει μία επιπλέον εβδομάδα για την κατάθεση τροπολογιών. Γιατί είναι σημαντικό ναι με να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, αλλά να υπάρχει και συμφωνία μεταξύ μας στα βασικά σημεία βλέπω ότι ήδη κάποιοι συνάδελφοι βλέπετε ήδη τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή πώς μπορούμε να διαπραγματευτούμε για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, όπως είπε ο κύριος Βλάζα. Καλά, ας βάλουμε κάποια θέματα επιτάπητος ήδη τώρα ως αφετηρία, να δούμε ποιες είναι οι αρχές, ποιες είναι οι βασικές μας ιδέες. Και μπορούμε να φτιάξουμε ένα πακέτο μετά. Εγώ είμαι αισιόδοξο είμαι θετικός. Μπορούμε να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα. Πράγματι, η πιστοποίηση, το accreditation θα τα διευκρινίσουμε. Και φυσικά όλα έχουν να κάνουν και με τον δημοσιονομικό κανονισμό που είναι σε εξέλιξη η σχετική επεξεργασία. Ίσως καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Θα πρέπει να δεχθούμε και κάποια πράγματα. πώς θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες των κρατών μελών, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, όλα αυτά είναι αναπόσπαστα κομμάτια αυτού του νέου κοινού συστήματος. Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά τώρα που είπατε για το κοινοτικό τα λοιπά, Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα συζητηθούν. Και το έχουμε ξανασυζητήσει άλλωστε αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά το αποθεματικό επιδόσεων, performance reserve. Δεν το θέλετε, ας μην καθίσουμε και εμείς να ασχοληθούμε τελικά με αυτό, δεν κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες διαδικασίες. Μπορεί να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών πολύ καλύτερος προγραμματισμός για την ανάπτυξη και για επενδύσεις σε τομείς που ενδυναμώνουν τα βασικά θεματικά, τους βασικούς θεματικούς στόχους. Με κρίση πλέον. Μην επανέρχεστε με τις προτάσεις σας. Δίνουμε σαφή μηνύματα στο Κοινοβούλιο. Και σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, ήταν σαφής θέση μας και εμένουμε σε αυτήν. Mr. President, maybe can... Δεν ξέρω αν η Κωνσταντζε μπορεί να πάρει το λόγο για να πει έτσι και αυτή την απόψή τη. Βεβαίω λέει ο πρόεδρος. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλο πάντων ναι, θα τη δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Λάμπερτ. Όχι, κάποιες παρατήρησει επιτρέψτε μου για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Αυτά εν μέρη περιλαμβάνονται στις τροπολογίες μας τα σχόλια που κάνατε για θέματα του performance reserve, για το ΦΠΑ, για τους εμπειρογνώμονες ε, συνέργειας και ρεσιμότητα εξάντε και στη σχέση της με την περιφερειακή πολιτική. Όλα αυτά τα έχουμε συμπεριλάβει στις τροπολογίες μας όντως. Τώρα, για το θέμα της πιστοποίησης και για το κλείσιμο των λογαριασμών. Να σας πω το εξής. Ε, εξαρτώμαστε από το δημοσιονομικό κανονισμό που βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας και διαπραγμάτευσης σήμερα. Άρα, συνάδελφοι, σας παρακαλώ μην κάνετε τροπολογίες για το θέμα αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είμαστε σε θέση να το κοιτάξουμε από μόνοι μας θέμα αυτό. Σε κάποια θέματα, όπως το θέμα της υπηρεσίας πιστοποίησης, εξαρτώμαστε από τις αποφάσεις για τον δημοσιονομικό κανονισμό και θα πρέπει μετά να κοιτάξουμε πού έχουμε περιθώριο ελιγμού για να αλλάξουμε κάποια ζητήματα ή όχι. Και το ίδιο θα ήθελα να πω ότι ισχύει αν υπάρχουν προτάσεις όντως για απλοποίηση, εμείς ε, ως εισηγητές ε, κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις για θέματα τέτοια απλούστευσης και είπαμε στους συναδέλφους αν υπάρχουν κάποιες δυνατότητες να υποβάλουμε τέτοιες προτάσεις. Κοιτάξτε, ομολογώ ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να απλοποιηθεί ένας τόσο σύνθετος μηχανισμός, γιατί αφενός ε, ε, όταν αλλάζουμε κάτι σε ένα τομέα, αυτό επηρεάζει ε, πάρα πολλούς άλλους τομείς και πολλοί αντιδρούν, ξέρετε. Και αυτό να το λάβουμε υπόψη στη συζήτηση αυτή. Ποιες είναι οι συνέπειες σε κάθε περίπτωση. Αλλά ασφαλώς αν υπάρχουν ε, έξυπνες τροπολογίες για την απλοποίηση της διαδικασίας, ευχαρίστως να τις λάβουμε και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο λόγια να πω για αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφαιρέσαμε τα key actions, τις κύριες δράσεις, γιατί δεν υπήρχε καμία αναφορά με τον Γενικό Κανονισμό. Δεν υπήρχε αναφορά για το τι ήταν. Αν ε, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι έξυπνο να μας πει, ασφαλώς θα τον υποστηρίξουμε. Αλλά γίνονται εντατικός διάλογος για το θέμα αυτό και για το θέμα του Performance Reserve. Φυσικά, η κατεύθυνση της ε, πολιτικής συνοχής θα πρέπει να είναι στα αποτελέσματα. Όχι μόνο να δημιουργούμε αριθμητικά στοιχεία, αριθμούς, νούμερα, αλλά να έχουμε και να πετυχαίνουμε και αποτελέσματα. Αυτό όλους μας συμφέρει. Και ο τρόπος που υπολογίζεται όμως το performance reserve δεν θεωρώ ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να το πετύχουμε αυτό. Αν έχουμε κάποια ε, ευφυή ιδέα και πρόταση για το θέμα αυτό, να τη συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να το θέσουμε και πριν την ψηφοφορία, όπως είπε και ο Γιάννη προηγουμένως. Βρισκόμαστε στην αρχή των διαπραγματεύσεων, των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι στον δρόμο για την μελλοντική πολιτική συνοχή θα πρέπει όλοι να κινηθούν και να συμμετάσχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου η πολιτική συνοχής να λάβει αυτή την, τον προσανατολισμό προς το μέλλον. Ε, μία κουβέντα να πω ακόμα, μιλώντας για συμβάσεις εταιρικής σχέσης, να μιλάτε για συμβάσεις εταιρικές εταιρική ε, εταιρικής να μην μιλάμε για συμφωνίες ε, εταιρική σχέση, γιατί θέλουμε να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα αυτέ τι συμβάσει και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και στις συζητήσεις με το Συμβούλιο, γιατί θέλουμε να συμπεριληφθούν και οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές, το που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις συμβάσεις αυτές εταιρικής σχέσης. Άρα, αυτό να διευκρινίζεται και σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Θα, είμαστε, θα σας ήμασταν ιδιαίτερα ευγνώμονε Ευχαριστώ. Κορνέλια, αν και δεν έχουμε χρόνο, 10 λεπτά. Ναι, μία ερώτηση θέλω να κάνω σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση και το κλείσιμο των λογαριασμών που με βρίσκουν αντίθετη. Είναι έξυπνο η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να μην πει τίποτα, να μην κάνει τίποτα. Να μην ψηφίσει καν ότι δεν του θέλει αυτό το πράγμα. Πώς θα μεταφερθεί το μήνυμά μας, τι άλλη ευκαιρία έχουμε για να αμυνθούμε κατά του μέτρου αυτού, γιατί πραγματικά είναι άσχημα τα στοιχεία αυτά. Το να μην κάνουμε τίποτα... Δεν μου φαίνεται σκόπιμο. Από τακτικής άποψης δηλαδή ενίσταμε. Κορνέλια, πολύ λυπάμαι, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας για το Financial Regulation έκθεση Γκρέσλε ο, πλειοψηφικά υπερψηφίστηκε το Κοινοβούλιο. Βρίσκεται σε διαδικασία συναπόφαση της διαπραγματεύση με το Συμβούλιο. Και το άρθρο 56 είναι ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά την ε, αρχή πιστοποίηση. και το Κοινοβούλιο είναι αυτό που επέμεινε για την αρχή αυτή πιστοποίηση, όχι το Συμβούλιο. Αυτή την απόφαση έλαβε το Κοινοβούλιο και πολύ απλά έχουμε καθυστερήσει. Δεν μπορούμε ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, των υστέρων να θέλουμε να αλλάξουμε την απόφασή μας. Και όπως σας είπα, στο διτακτικό του κανονισμού αναφέρεται ότι ο... η αρχή πιστοποίησης έχει να κάνει με το άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού είναι ομοθεσία, τι να σας πω, και εμένα με δεσμεύει. Δεν μπορώ να έρχομαι εκ των υστέρων και να αμφισβητώ εθελούσια τέτοια πράγματα. Αν δεν το θέλαμε, έπρεπε πολύ πολύ νωρίτερα να είχαμε σκεφτεί ποια θα ήταν, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στην περιφερειακή πολιτική. Τώρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε να συζητήσουμε ίσως με την κυρία Γκρέσλα μήπως θα μπορούσαμε να πετύχουμε ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο, αν και αυτό πρέπει να σας πω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα, αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα ε, τις για το γενικό κανονισμό. Να πω ότι συνάδελφοι η 7η Ιουνίου είναι η καταλεκτική ημερομηνία για κατάθεση τροπολογιών για το γενικό κανονισμό μέχρι 31 Μαΐου. 7 ε, Μαΐου για το CSF. Να επαναλάβω ότι δεν ακολουθούμε τις κανονικές διαδικασίες, ακολουθούμε μια ειδική διαδικασία, όπως ξέρετε, η οποία προτάθηκε από τη Γραμματεία και οι οδηγίες θα σας αποσταλούν σύντομα από τη γραμματεία όσοι θέλετε να καταθέσετε τροπολογίες για το CSF και δεν ξέρετε πώς να το κάνετε, πριν τις υποβάλλετε, ε, ε επικοινωνήστε με τη γραμματεία και να περάσουμε στην έκθεση του Γιώχημ Τσέλερ. Γιώχημ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αλλάξατε και τη σειρά των σημείων στην ημερήσια διάταξη για να μιλήσουμε και για το σχέδιο κανονισμού για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας. Θα είμαι αρκετά σύντομος. Τρεις φορές στην Επιτροπή άλλωστε έχουμε συζητήσει τον τροποποιημένο κανονισμό, την πρόταση κανονισμού και στο μεταξύ έγινε και μια ακρόαση από το, την ομάδα του ΕΛΚ για το θέμα ότι εξή, ε, ότι η, Ευρω... Επιτροπή των Περιφερειών έχει εκφράσει σχετικέ απόψεις ε, και πάρα, πολύ πάρα πολλές περιφέρειες ε, προγραμματίζουν νέους ομίλους εδαφικής συνεργασίας και φαίνεται ότι τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο ο Ευρωπαϊκός Ομίλος Ανταφικής Συνεργασίας θα αποτελέσει το νομικό μέσο για την οργάνωση της διασυνοριακής συνεργασίας. Ο κανονισμός ο οποίος μας προτείνεται στο σημείο αυτό, σε αντίθεση με τις άλλες ε, δομές κανονισμών, έχει το εξής ε, προτέρημα. Δεν είναι καινούριος ε, κανονισμός βασίζεται στον κανονισμό του 2006. Τον διευρύνει και τον το τροποποιεί. Συμπεριλαμβάνονται τα σχόλια των περιφερειών που ήδη εργάζονται με Ευρωπαϊκούς Ομίλου Οδακτική Συνεργασία. Και διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των εταίρων που θα συμπεριλαμβάνονται. Για παράδειγμα, οι δημόσιες επιχειρήσεις στο μέλλον θα μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Ομίλου Δαφικής Συνεργασίας. Θα μπορούν να υπάρχουν διμερεί όμιλοι ε, διασυνοριακής συνεργασίας, δηλαδή ε, μεταξύ ενός μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός μη μέλους. Και επίσης θέλουμε να μην είναι μόνο αυτό θέμα περιφερειακής πολιτικής και διαρθρωτικών ταμείων, αλλά και οι όμιλοι ταφικής συνεργασίας να χρησιμοποιούνται και σε άλλο τομεί πολιτικής σημασίας ε, στο σύντημα ορίζοντας 2020 ε, και το καθεξής. Θέλουμε ως νομικές οντότητες η Ευρωπαϊκή Όμιλη Ταφικής Συνεργασίας να μπορούν να συμμετέχουν σε πολιτικούς τομείς και σημαντικό είναι το εξής. Οι πολλαπλές αρχές πιστοποίησης που υπάρχουν ε, σε κάθε κράτος μέλος να περιοριστούν αριθμητικά προκειμένου όσοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο όμιλο στο μέλλον να έχουν να κάνουν με μία υπηρεσία πιστοποίησης ανά κράτος μέλος και να μην υπάρχουν να μην ε, χρειάζεται να απευθύνονται σε πάρα πολλές υπηρεσίες. Τώρα, η μεταφορά σε εθνική νομοθεσία. Αυτό είναι το επιθυμητό. Και αυτό και συστήνουμε κατεπηγόντως. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού έχουμε καταλήξει σε μια γενική συνένεση. Λίγο πιο αντιστακτικό είναι το Συμβούλιο δυστυχώς σε ό,τι αφορά την τροποποίηση του κανονισμού. Δεν καταφέραμε ακόμη να μάθουμε ποια είναι η επί της αρχής τοποθέτηση του Συμβουλίου. Η, ως νομική ως ε, οντότητες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατανέμουν και αρμοδιότητες. Η Ευρωπαϊκή Όμιλη Δαφική Συνεργασία. Κάποιοι φοβούνται στα κράτη-μέλη ότι με τον τρόπο αυτό μεταφέρονται και δίδονται αρμοδιότητες. Εμείς δεν συμφωνούμε. Ελπίζω μέσω της μελλοντική συζήτησης με το Συμβούλιο να καθυσυχαστούν και να διασκεδαστούν οι ανησυχίες αυτές, προκειμένου οι όμιλοι εδαφικής συνεργασίας στην επόμενη προγραμματική περίοδο να αναπτυχθούν πλήρως ως μέσο διασυνοριακής περιφερειακής ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Very much. Ευχαριστώ πολύ η Μόνικα Σμόλκοβα. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. θα πρέπει οπωσδήποτε να εκφράσω την εκτίμησή μου για την εργασία του κυρίου Τζέλερ. Εξαιρετικό το έγγραφο εργασίας και οι τροπολογίες ιδιαίτερα χρήσιμες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του κανονισμού, δηλαδή ε, η δημιουργία αυτών των ομίλων εδαφικής συνεργασίας. Όταν η Κομισιόν υπέβαλε την πρότασή της, ξεκίνησε μια διαδικασία διαβουλεύσεων και διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς ε, έλαβαν μέρος. Ο εισηγητής υπέβαλε μόνο, και αυτό το βάζω μετά σε εισαγωγικά, 23 τροπολογίες. Θα ήθελα να αναφέρω μερικές από αυτές τις τροπολογίες. Υπαριθμόν ένα που είναι πάρα πολύ καλή και αφορά το ποιες επιχειρήσεις θα πρέπει να εμπλακούν. Αυτές οι οποίες παρέχουν ε, ε, υπηρεσίες και είναι γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης, μου αρέσει και η τροπολογία 5 που αναφέρεται στην διασυνοριακή συνεργασία και ο εισηγητής ε, αναφέρθηκε σε αυτό και στην, ε, στην, ε, στο προήμιο, στην εισαγωγή. Η τροπολογία 6 ίσως είναι λίγο αμφιλεγόμενη, είχα κάποιες ε, κάποιες αμφιβολίες αλλά όταν τελικά ε, τοποθέτησα κατά κάποιο τρόπο την τροπολογία αυτή στο ευρύτερο πλαίσιο και έλαβα υπόψη μου και τις ε, πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές τελικά θεωρώ ότι και η τροπολογία 6 μια χαρά είναι. Όσοι δεν την διάβασαν η τροπολογία 6 λέει ότι αυτοί οι όμιλοι θα πρέπει να θεωρούνται ε, εργαλείο καθολικής ε, συνεργασίας και θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για κάθε είδους ε, χρηματοδότησης. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου επ' αυτού. Εν συμφωνώ απολύτως με την τροπολογία 8 καθώς επίσης και τις άλλες τροπολογίες οι οποίες έχουν στόχο την αποσαφήνιση ή την απλούστευση του κειμένου. Νομίζω ότι μένουν τρει-τέσσερι τροπολογίε για τι οποίε μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση, αλλά είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να τη στηρίξουμε έτσι ώστε να απλουστευτεί περαιτέρω το κείμενο. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα τούτο θα γίνει ε, ιδιαίτερα καλό και για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ναι, ε, Πρέπει να πω ότι είμαι ευτυχής με την έκθεση αυτή και με, την, ε, με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των προτάσεών μας αντικατοπτρίζονται στο κείμενο το οποίο μας έχει υποβληθεί. Ε, είναι καλό όλα αυτά που λέγονται για απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ, Ε, καθώς επίσης ε, ε, και όσον αφορά και τους εργαζόμενους και τα λοιπά. Και αργότερα θα επανέλθω. Πρόεδρος, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Διαφορετικά θα δώσουμε αμέσως το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος είναι ο εκπρόσωπος. Δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Εντάξει. Είναι λίγες οι τροπολογίες φαίνεται και δεν αποτελούν κίνητρο. David, as much time as Ντέιβιντ, ε, έχει όσο χρόνο χρειάζεσαι. Δεν πήραν το λόγο πολύ συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ σε αυτή τη φάση. Να υπογραμμίσω μονάχα ότι η Κομισιόν εκτιμά ιδιαίτερο στη θέση της Επιτροπής, κυρίως δε του εισηγητού, ο οποίος κατανόησε την ουσία και την βάση αυτού του τροποποιητικού κανονισμού. Ε, δεν θα σας δώσω αυτή τη στιγμή ε, οποιαδήποτε, ε, οποιοδήποτε δεν θα κάνω κήρυγμα όσον αφορά ε, τις τροπολογίες και που έγιναν δεκτές και όχι. Πάντως χαίρομαι που έγινε κατανοητός ο στόχος της Επιτροπής όσον αφορά τις ε, άλλες τροπολογίες εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν τροπολογίες τις οποίες θεωρούμε βοηθητικές έτσι ώστε να απλουστευτεί περαιτέρω ή να εξηγηθεί καλύτερα το περιεχόμενο εκεί που εμείς δεν ε, καταφέραμε να εξηγήσουμε καλά ε, το κείμενο πριν από μερικούς μήνες όταν το υποβάλαμε ας πούμε. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η αναφορά στις δημόσιες προμήθειες ε, εδώ ίσως χρειαζόταν κάποια επεξηγηματική σημείωση όντως ε, μπορούμε κάλλιστα να βασιστούμε στην ε, νομολογία μια και δεν το είχαμε κάνει μέχρι τώρα. Επίσης σε σχέση με το μητρό του των ομίλων εδαφικής συνεργασίας που θα πρέπει να κρατάει η, περιοχή, συγγνώμη, η Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, και χαιρόμαστε που θέλουν να στηρίξουν και εκείνη αυτή την τροπολογία. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που έχουν την ίδια έτσι, ακολουθούν την ίδια απώλεια. Δεν θέλω να χαλάσω αυτή την ωραία ατμόσφαιρα, λέει ο μιλητής. Ε, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες ε, με τις οποίες δυσκολευόμαστε όσον αφορά τη νομική τους βάση κυρίως. Ε, κυρίως ε, τροπολογίες οι οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις που αφορούν άλλα πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας. Δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν δηλαδή διατάξεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει αποδεκτές και αποτελούν ενωσιακή νομοθεσία αυτές οι προτάσεις τροποποίησης, ε, έστω και αν καταλαβαίνουμε το κίνητρο τους ε, και το πνεύμα το οποίο αποτελεί την βάση τους, ε, παρόλα αυτά, επειδή εμπλέκονται νομικά ζητήματα, δεν μπορούμε να τις δεχτούμε. Ευχαριστώ πολύ έχουμε το χρόνο να ακούσουμε και τις νομικές και τη νομική επιχειρηματολογία. Θέλετε να μας πείτε τώρα είναι σημαντικό για τον εισηγητή να ακούσει και τη νομική αιτιολόγηση. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε ο υπάρχουν κάποια νομικά προβλήματα σε ό,τι αφορά κάποιες από τις προτάσεις που πίπτουν σε τέσσερις κατηγορίες. Όπως ανέφερα ήδη, υπάρχουν ε, κάποιες προτινόμενες τηλεογικές σκέψεις ε, οι οποίες ε, υποδεικνύουν άλλους πολιτικούς τομείς και εκεί θεωρούμε ότι δεν είναι σωστός ε, χώρος ο κανονισμός αυτός να αναφέρονται άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές όπως το είπα για παράδειγμα το ENI. Αλλά προσπαθούμε με τις άλλες υπηρεσίες να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να ληφθεί υπόψη και το θέμα αυτό. Ένα άλλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο ε, αλλάζουν, τροποποιούνται οι κανονισμοί. Σε ό,τι αφορά τροπολογίες 2 ε, και 4. Γίνεται αναφορά στο άρθρο, άρα το άρθρο αποτυπώνει την αιτηλογική σκέψη που προετοιμάζει το διδακτικό Άρα αυτό που ρυθμίζεται, που θέλουμε να ρυθμίσουμε, θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στην αιτιολογική σκέψη και όχι μόνο να αναφέρεται στο διδακτικό στο άρθρο. Η αναφορά τώρα στην πρόταση 20 για το άρθρο 16 του υφιστάμενου κανονισμού. Δεν είναι σαφής, σαφές το τι ακριβώς προτείνεται. Τι αλλάζει μία παράγραφος, θέλετε να προσταθεί ή μία υποπαράγραφος, μία τρίτη ομάδα τώρα. Έχει να κάνει με την σχέση για τις προτάσεις αλλαγών αντιλογικών σκέψεων και των αντίστοιχων άρθρων που δεν συνάδουν. Για παράδειγμα, στην ε, τροπολογία 10 προτείνεται μία τελογική σκέψη η οποία όμως δεν συνοδεύεται από αλλαγή σε κάποιο άρθρο. Αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσον η πλατφόρμα της, Ευρω... της Επιτροπής της Προεδριών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην Ευρώπη του 2020. Αντιστρόφως, οι προτάσεις ε, για νέες ε, προδιαγραφές στον κανονισμό στη τροπολογία 2021 και 2023 δεν συνοδεύονται από τη λογική σκέψη. Δεν υπάρχει προετοιμασία δηλαδή σε τη λογική σκέψη. Τέταρτη ομάδα, τροπολογίες. για τις οποίες δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε καταλάβει ακριβώς τι εννοείται. Όπως οι 8 και οι 17, για παράδειγμα, δυνατότητα των ομίλων ταυτικής συνεργασίας να συνάπτουν συμβάσεις με άλλες νομικές οντότητες. Επειδή είναι νομική οντότητα ο ομίλος ταυτικής συνεργασίας, αυτό ασφαλώς και ισχύει. Δεν χρειάζεται, θεωρούμε, να τονιστεί ιδιαίτερα εκ νέου στην τροπολογία 9 τώρα. Αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το εφαρμόσιμο δίκαιο να ορίζεται στη συμφωνία. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να αναφέρεται για παράδειγμα ότι για αυτό τον όμιλο δεδική συνεργασία ισχύει το γαλλικό δίκαιο. Αυτό έτσι κι αλλιώ είναι σαφέ. Υπάρχει μια λίστα συγκεκριμένων προδιαγραφών σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τις δραστηριότητες ενός ομίλου δαφικής συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό τμήμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και σε μια τη σκέψη, γιατί θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια για το ποιοι κανόνες ισχύουν για το προσωπικό ενός ομίλου ταφικής συνεργασίας. Τροπολογία 19 τώρα. Θέλει εκ νέου να διαγράψει την περίπτωση περιορισμένη ευθύνη ε, σε ομίλους οδαφικής συνεργασίας. Κοιτάξτε, ξέρουμε και τις ε, ε, εταιρείε περιορισμένη ευθύνη. Από το περιορισμένη ευθύνη προκύπτει αυτή η περιορισμένη ευθύνη των ε, επιχειρήσεων. Αυτό ε, προειδοποιεί κατά κάποιο τρόπο τους εταίρους της νομικής αυτής οντότητας σε κάθε περίπτωση. Τώρα, για την τροπολογία 20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πει στην Επιτροπή των Περιφερειών τι θα κάνει με την πλατφόρμα της. Αυτό δεν μας βοηθάει. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα πρέπει να ξέρει τι θα κάνει με την πλατφόρμα που έχει αναπτύξει και που λειτουργεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλά θα ακολουθήσει. Τέλος, στην τροπολογία 14 προτείνεται η σύμβαση ε, και σύναψη και ιδρύση ενός ομίλου ενταφικής συνεργασίας να δημοσιοποιείται σε όλες τις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα λόγω των 23 επίσημων γλωσσών. Γι' αυτό αυτό που προβλέπεται στην, στον παρόν κανονισμό είναι να δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ίδρυση ενός ομίλου ενταφικής συνεργασίας και όποιος επιθυμεί σε όλη την Ευρώπη μπορεί να συμβουλεύεται τα απαραίτητα έγγραφα. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να τα συζητήσει όλα αυτά και λεπτομερέστερα με τον εισηγητή. Uh, uh, Προεδρο, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Δεν ξέρω αν ο Ιωχήμ θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που μου προτείνετε να συζητήσουμε. Ωστόσο, κάποια από τα επιχειρήματα, από τις σκέψεις που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, με βρίσκουν σύμφωνο. Δεν τα καταλαβαίνω. Όταν μιλάτε για σύγχυση και αντίθεση με άλλους ε, τομείς της πολιτικής σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία, την ΕΠΑ, τη σύμβαση σε ΕΠΑ. Αυτή ήταν η πρόθεση να συμπεριληφθούν, να μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλοι πολιτικοί τομείς. Γιατί αν δίνουμε στην δυνατότητα σε έναν όμιλο εδαφική συνεργασία ε, να συνεργαστεί και με τρίτα κράτη, είναι συνήθω ποια κράτη είναι αυτά, τα κράτη γειτονία. Άρα ουσιαστικά εμπεριέχονται συνήθω στην ε, πολιτική γειτονία. Άρα αυτό καλό είναι και οδηγεί στην δικτύωση των πολιτικών και σε μια συνοπτική ε, και συνεκτική ε, προσέγγιση. Για την τροπολογία 20, για την Επιτροπή των Περιφερειών υπάρχει και μία δεύτερη φράση για το λόγο για τον οποίο θέλουμε να συμπεριληφθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συμμετέχει στην πλατφόρμα αυτή για να πετύχουμε καλύτερη επικέντρωση στους συγκεκριμένους πολιτικούς τομείς που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, για να επικεντρωθούμε και να μειωθεί το θέμα, αν θέλετε, σε θέματα μόνο ε, της αντικής πολιτικής, αλλά να υπάρχει και μια πιο ευρύτερη προσέγγιση. Αυτό αποτέλεσε επιθυμία και των περιφερειών. Ε, κοιτάξτε, εγώ με χαρά θα συνεχίσω τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ε, από ό,τι φαίνεται μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. 31η Μαΐου η προβολή, συγγνώμη, προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Δεν υπάρχει αλλαγή ε, όσον αφορά το ωράριο την ώρα μάλλον που θα έρθει ο Επίτροπος. Δεν έχουμε, ε, έχουμε λοιπόν 10 λεπτά μπροστά μας. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να θίξετε εντωμεταξύ. Όχι, από ό,τι φαίνεται όχι. Επομένως θα περιμένουμε 10 λεπτά και θα διακόψουμε περιμένοντας στις 11 τον Επίτροπο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνάντηση με τον Επίτροπο ακριβώς στις 11. Και επίσης να θυμίσω στους συναδέλφους ότι τρεις η ώρα θα έχουμε από κοινού με την Ήτρε μια πάρα πολύ σημαντική ακρόαση ε, όσον αφορά την πολιτική συνοχή και τον ορίζοντα 2020. Μετά θα έχουμε ψηφοφορίες. Γι' αυτό σας παρακαλώ να έρθετε και το απόγευμα. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξαναρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Έχει έρθει εδώ ο Επίτροπος. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Γιωχάνες Χάν Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε την μια μισή ώρα που έχουμε ε, μαζί με τον Επίτροπο έτσι ώστε να αποσαφηνίσουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε στο μυαλό μας. Όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν ε, είναι καλοδεχούμενες οι ερωτήσεις τους ε, έτσι ώστε ό,τι έχουν στο νου τους να τα απαντήσει ο Επίτροπος. Κύριε Επίτροπο έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μιλήσω εδώ στην Επιτροπή σας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συγκυρία για όλους μας και ιδιαίτερο για εμένα σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της ε, περιφερειακής πολιτικής και για... θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας ε, την ε, κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Βλέπουμε και ζούμε, διανύουμε μία περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάμε για επιπλέον κίνητρα και ξεχνάμε ότι με τα μία ταμεία μας δίνουν ήδη ένα υφιστάμενο μέσο τέτοιων κινήτρων. Ο πρόεδρος Μπαρόσο την προηγούμενη εβδομάδα, εβδομάδα μίλησε και είπε ότι η μεταρρύθμιση πάει χέρι με χέρι με τις επενδύσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και στις νέες θέσεις εργασίας. Μίλησα για ανάπτυξη. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν ανοιχτά ποια μέσα θέλουμε να ενισχύσουμε και πώς. Αυτή την ορμή θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής και στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου. Χρειαζόμαστε γρήγορες ε, αποφάσεις στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα για τα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία θα πρέπει να βεβαιωθούν μέχρι τα τέλη του 2020. Να συγχαρώ την Επιτροπή σας για την ε, πολύ γρήγορη διαβούλευση σας ε, για την... Ε, μάλλον, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω και το Συμβούλιο να σημειώσει καλή πρόοδο, να σας παρουσιάσω πώς έχουν τα πράγματα και ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής και πώς τοποθετούμαστε έναντι της στάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποια ζητήματα στρατηγικού προγραμματισμού, ε, αιρεσιμότητας 60 και μέσων απλούστευσης συζητήθηκαν προκαταρτικά. Φυσικά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί εφόσον δεν έχει αποφασιστεί το συνολικό πακέτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποστηρίζει ούτε το Συμβούλιο ούτε το Κοινοβούλιο στην φάση αυτή, αλλά ε, βλέπει το ρόλο της ως ρόλο διαμεσολαβητή και είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχουν οποιασδήποτε συμφωνίες με έναν από τους δύο νομοθέτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποστηρίζει την νομοθετική της πρόταση. Κατά το παρελθόν πάντα υπήρχαν ερωτήσεις για τα negotiating boxes όπως αποκαλούνται μέσα της Προεδρίας του Συμβουλίου για τις ε, δομές και την διάρθρωση της συζήτησης στο ιστορικό του Συμβουλίου. Αυτό το αποδέχεται το Κοινοβούλιο, το, η Επιτροπή. Αλλά δεν επηρεάζεται έτσι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, τρία σημεία θα ήθελα να αναφέρω που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για όλα τα διευθυντικά ταμεία. Είναι πολύ σημαντικό για το συνολικό πλαίσιο της πρότασης μεταρρύθμισης. Ξέρω ότι εξ αρχής ήταν διαφορετικές οι θέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των δύο νομοθετών. Αφετέρου σε ό,τι αφορά το νομοθετικό χαρακτήρα, το νομικό χαρακτήρα του πλαισίου αυτού, αλλά ξέρω ότι συμφωνούμε ότι το μέσο αυτό είναι απαραίτητο. Το θέμα είναι η ουσία της πρότασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πρόθυμη να μιλήσει με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου για ένα παράρτημα, το οποίο θα αποτελέσει, μάλλον δεν θα ε, προκαλέσει ε, ακύρωση της ε, πράξης τις εκτελεστικής πράξεις, Θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα του παρατήματος και της, ε, του διαχωρισμού των θεμάτων, προκειμένου να καταλήξουμε σε μία συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από κάποιες εβδομάδες υπέβαλε μία πρόταση για την αλλαγή του κώδικα αντιντολογίας σε ό,τι αφορά τη συμβάση συντηρική σχέσης και είμαι βέβαιος ότι η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το πόσο δεσμευτική θα είναι η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δυστυχώς πρέπει να σας αναφέρω ότι από πλευρά Συμβουλίου υπάρχει κάποιος δισταγμός. Καλό λοιπόν το Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή κρατικών και μη κρατικών οντοτήτων, σε ό,τι αφορά τη θεματική επικέντρωση τώρα, κυρίε και κύριοι. Η τρέχουσα συζήτηση για τη σωστή ισορροπία μεταξύ μέτρων ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη καταδεικνύει το εξής, ότι θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε πιο εντατικά πώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα περιορισμένα μέσα. Παρακολουθώ τις συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τη συζήτηση επικέντρωση κατά ε, της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανοιχτή για τέτοιες ε, ιδέες εφόσον δεν διακυβεύεται η βασική αρχή της επικέντρωσης. Αν η ευελιξία όμως σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να συγκεντρώσουμε μία κρίσιμη μάσα, μάζα και να συμβάλλουμε στην εφαρμογή της ε, πολιτικής ε, ανάπτυξης και ενοποίησης και ενσωμάτωσης. Και στην περίπτωση αυτή η, ευρωπαϊκή, η μεταρρύθμιση αυτή θα έχει αποτύχησαν ένα από τους βασικούς στόχους της. Αν θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή είναι πολιτική ανάπτυξη, θα πρέπει να επενδύσουμε εκεί πέρα που πραγματικά υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης και εκεί που θα κρυθεί ο ανταγωνισμός ο, ο παγκόσμιος τα επόμενα χρόνια στην ε, δυναμική οντομία των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων, στην ε, καμπή της ενεργειακής ε, παραγωγής, στην επένδυση σε πράσινες και μπλε τεχνολογίες αλλά και σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Αν επιτρέψουμε οι προτεραιότητες αυτές να αποδυναμωθούν ή να διευρύνονται διαρκώς, το κίνητρο ανάπτυξης για τις περιφέρειές μας και για τις επιχειρήσεις μας θα είναι πολύ περιορισμένο και προκειμένου κυρίες και κύριοι να μην αποδυναμωθεί η αποδοχή, η αναγνώριση της πολιτικής μας, θα πρέπει στο μέλλον να την ενισχύσουμε, να την κάνουμε πιο ορατή, να δώσουμε πολιτικά κίνητρα. Ας συζητήσουμε λοιπόν με ανοιχτό πνεύμα πώς ε, μπορούμε να επιτρέψουμε στις περιφέρειες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκριθούν στις σχετικές ε, ανάγκες, χωρίς να διακυβεύονται οι γενικότεροι στόχοι της στρατηγικής 2020 σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Η Ευρώπη χρειάζεται την ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίες. Αν συνεργαστούμε για μια βιώσιμη πολιτική επένδυσης για την Ευρώπη, για τις περιφερειές μας, θα σας παρακαλούσα αυτό να μην το ξεχνάμε, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο, όχι μόνο για την επιτυχία της πολιτικής, αλλά για την επιτυχή έξοδο της Ευρώπης από την πολύ δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση για να μην την αποκαλέσω κρίση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ξεκινήσουμε ως συνήθως με τους συντονιστές. Ο Λάμπερτ Φανίλ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ, κύριε Επίτροπε, ιδίως αυτή τη χρονική στιγμή, πάρα πολύ επίκαιρη η επίσκεψή σας. Είναι πολλοί συναδελφοί θέλουν το λόγο. Ας έχουμε λοιπόν μια ανοιχτή επικοινωνία. Ίσως το σημαντικότερο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να προσφέρει πραγματικά η περιφερειακή ανάπτυξη και όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για την ενίσχυση της οικονομίας μας, πώς μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην ένταξη των πολιτών. Μήπως ε, είμαστε πολύ συγκρατημένοι και επιφυλακτικοί. Μήπως πιστεύουμε ότι όλοι στις ε, χώρες μας, στις διαπραγματεύσεις, δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς ε, τα ωφέλη που μπορεί να παράσχει η περιφερική πολιτική. Γιατί κάνω αυτά τα ερωτήματα. Ίσως να μην συμμετέχω στις σωστές συζητήσει, αλλά σε κάποια τραπέζια που έχω καθίσει ακούω πολλές φορές ότι ναι όλα αυτά είναι πολιτική, οι πόροι αυτοί δεν χρησιμοποιούνται, πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές εντελώς κτλ. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική συμμαχία, αν θέλετε, μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου, που πρέπει να αξιοποιήσουμε για να διευκρινίσουμε το πώς μπορεί να συνεισφέρει η περιφερειακή ανάπτυξη ε, ε, στην ανάπτυξη γενικότερα και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το περιβάλλον. Τέτοιου είδους ερωτήματα δεν αφορούν μόνο το Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξη, αλλά και το Ταμείο συνοχή και το Κοινωνικό Ταμείο. Ίσως λοιπόν πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Δεύτερον, μη σε πιστώσεις. Θα μπορούσατε να δώσετε σαφή στοιχεία για την κατάσταση, γιατί πολλοί δεν κατανοούν ακριβώς τι γίνεται νη συν 2, νη συν 3, πιστός πληρωμών. Είναι πράγματα που δεν τα κατανοεί ο κόσμος ε, και όταν υπάρχουν ε, περικοπές σε εθνικό επίπεδο, ε, είναι δύσκολο να πούμε ότι χρειαζόμαστε στην Ευρώπη περισσότερα χρήματα και δι για την συνοχή. Και έχουμε και τη συζήτηση του 2013. Μήπως θα έπρεπε αυτά τα στοιχεία, τα νούμερα να τα διευκρινίσουμε, είμαστε πιο άμεση απέναντι στον κόσμο. Επίσης πρέπει να πω ότι με χαροποίησε ιδιαίτερα αυτό που είπατε, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στις προτάσεις της. Δεν υπάρχουν συμφωνίες. Από ό,τι κατάλαβα δεν έχει ακόμα υπάρξει κάποια συμφωνία. Σε ό,τι αφορά το γενικό κανονισμό. δεν έχει γίνει κάποια ε, συμφωνία με τη Δανική Προεδρία. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον ε, στα περισσότερα ζητήματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις μετά την ψηφοφορία στις 9 Ιουλίου. Άρα έχουμε δυνατότητες. Δεν έχουν κλείσει κάποια κουτιά, δεν έχουν ολοκληρωθεί συζητήσεις για κάποια σκέλη των διαπραγματεύσεων. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα πλήρους συνομοθέτησης επί του συνόλου του πακέτου. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απεμπολίσουμε τις ευθύνες μας ή τις αρμοδιότητες που έχουμε. σε σχέση με κάποια διαπραγματευτικά κουτιά σε επίπεδο Συμβουλίου. Όπως είπατε και στην αρχή, πρέπει να έχουμε τη στήριξή σας, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό θα πρέπει να παραμείνει άθικτο. Είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα του Κοινοβουλίου. Είμαι βέβαιος ότι και οι συνάδελφοί μου θα σχολιάσουν. Ε, αυτά είχα να πω εγώ πάντως. Ευχαριστώ πολύ. Η Κωνσταντσε τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι συγητές ε, για τον κανονισμό για τα ταμεία έχουν καταθέσει τις προτάσεις μας και στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχή είναι καλή εξετάζοντας ε, το πού επιθυμούμε αλλαγές. Δεν είναι προς την κατεύθυνση επηρεασμού και αλλαγής του συνολικού μηχανισμού, ακόμα και αν υπάρχουν φυσικά σε κάποια σημεία διαφορετικές απόψεις μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις προτάσεις που μας έχετε καταθέσει. Μία ερώτηση φυσικά έχω να σας κάνω. Επίτροπε, ξέρετε ποιες είναι οι προτάσεις μας, ξέρετε τι περιλαμβάνεται στα negotiation boxes στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων λοιπόν. Αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι πώς εκτιμάτε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας. Πού μπορείτε να υποστηρίξετε το Κοινοβούλιο. Ο Λάμπερ ανέφερε το ερώτημα, το θέμα του ότι επιμένουμε στο δικαίωμα συναπόφασής μας. Ε, αυτό ασφαλώς ε, έχει άλλη διάσταση αν μας υποστηρίζετε και εσείς. Ε, δεν ξέρω όμως αν αυτό ισχύει. Πείτε μας. Και υπάρχουν και στοιχεία τα οποία συζητιώνται στο Συμβούλιο και θεωρώ ότι αξίζουν να υποστηριχθούν. Για παράδειγμα, η ιδέα για τα λειτουργικά προγράμματα και την διαίρεσή τους σε δύο τομείς για την πιο ευέλικτη διαμόρφωσή τους. Αυτά μου φαίνονται ενδιαφέροντα και σίγουρα μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής θα συζητηθούν το πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε τον κώδικα διοντολογίας. Θα κάνουμε και μια σχετική τροπολογία και θα υποστηρίξουμε την πρόταση αυτή. Είναι σαφές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που άκουσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτίθεται να συζητήσει θέματα παραδείγματος μαζί μας. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί νομίζω ότι τον ίδιο στόχο επιδιώκουμε με το Common Strategic Frame. Να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Φυσικά υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι δύσκολα. Performance Reserve, τα ακούσαμε και προηγουμένως, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα, multi-fund, προσβασιμότητα σε πολλαπλά ταμεία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία σίγουρα θα πρέπει εκτενώς να συζητηθούν. Ένα ωστόσο μου έκανε εντύπωση και σας παρακαλώ να το πω ξεκάθαρα. Ζήτησα από τους συναδέλφους στην Επιτροπή να θυμούνται γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει υποχωρήσεις και κάνει εκ των υστέρων και ε, συμφωνίες ε, με τα κρατημέλη και όχι συμβάσεις. Για πείτε μας, εμείς θέλουμε να υπάρχουν συμβάσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που θα συμμετέχουν, στις οποίες θα συμμετέχουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί αυτό το θέλουμε, θέλουμε να υποστηριχθούν. Μία διευκρίνηση λοιπόν για το ότι πραγματικά είναι συμφωνίες, ε, είναι συμβάσεις και όχι συμφωνίες. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική η κίνηση διαπραγματεύσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να καταλάβουν όλο και πιο πολύ στο Συμβούλιο ότι στην πολιτική ε, συνοχής θα βρουν μία πολιτική με την οποία μπορούν να ασκήσουν πολιτική επενδυτική και ανάπτυξης. Αυτό φαίνεται ότι φτάνει και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, βλέποντας πώς άλλαξε, για παράδειγμα, ο ευρωπαϊκός τύπος ε, τις τελευταίες εβδομάδες. Ε, αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική ανάπτυξης. Αυτό θα μπορούσε να μας δώσει τη δυνατότητα να προωθήσουμε το Κοινοβούλιο και την αξίωση του Κοινοβουλίου που είναι πιο υψηλή από τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαντάζομαι ότι θα μας υποστήριζε ενδεχομένω για τη σημασία της πολιτικής συνοχής πρόκειται να ε, αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και αν συνδεθεί με μια μεταρρυθμισμένη, σύγχρονη πολιτική συνοχή, νομίζω ότι με καλή συνείδηση θα μπορέσουμε να προτείνουμε ένα τέτοιο ισχυρό μέσο ανάπτυξη και ελπίζω να βρούμε έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε καλύτερα. of Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, λέει ο κ. Θα ήθελα όμως δύο λόγια να πω και να το υπογραμμίσω στον Επιτροπό. Πρώτα απ' όλα, η παρούσα κατάσταση, η υφιστάμενη κατάσταση που συνδέεται με το μέλλον. Το πρόβλημα είναι ότι στην Επιτροπή Προπολογισμών, γιατί είμαι και εγώ μέλος εκεί, συζητούμε το θέμα των αποθεματικών για τα επόμενα χρόνια. Και το πρόβλημα είναι ότι όσον αφορά τα χρήματα για την ε, συνοχή έχουμε λιγότερα, 5,5. Τα χρήματα λοιπόν δεν είναι πολύ καλά. Εάν βγάλουμε το μηχανισμό Connecting Europe, δεν μένουν και πάρα πολλά. Και βεβαίως ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Ενδεχομένω κάποιες χώρες θα ζητήσουν και για κάποια άλλα μείον στον υπολογισμό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος. Το πρώτο που πρέπει να υπογραμμίσω στον κύριο Χάν είναι το θέμα των ράλς ρέστα λικιντέ. Σύμφωνα με τον κύριο Λεβεντόφσκι, μπορεί να είναι ε, πολλά χρήματα, εκ των οποίων 70% αφορούν ε, την συνοχή. Και δεν καταλαβαίνουμε, τουλάχιστον εμείς ε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ενδεχομένως εδώ, ξέρουν καλύτερα, είναι πιο εξοικειωμένοι με την κατάσταση. Τα ΡΑΛ είναι τα χρήματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν εκταμιευτεί και δεν μπορούμε να βασιστούμε πάνω σε αυτά. Η άλλη γνώμη είναι διαφορετική, ότι όλα θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τελευταίο κέρμα. Θα ήθελα κάποια αποσαφήνιση. Γιατί έχουμε το πρόβλημα του 10 συν 2, 10 και 3. και βεβαίως τα χρήματα από το 2000 μέχρι το 2006 που θα μπουν στην συνοχή, που μπαίνουν στη συνοχή μέχρι τώρα, είναι πληρωμένα σωστά και υπάρχει αποθεματικό ή όχι. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι χρησιμοποιούμε αποθεματικά μέχρι το 2013, αλλά δεν είναι δυνατόν να πληρώσουμε 5 ε, δις τη στιγμή που η Επιτροπή δεν θα έχει δυνατότητα να τα πληρώσει αυτά μέχρι το Δεκέμβρη ε, ή θα πρέπει να μπουν την τελευταία στιγμή ως έσοδα στο 10 συν 2. Αυτή η ιδέα του να μπει περισσότερο μαθηματικό στην ε, ε, στην συνοχή, εμένα με αφήνει ιδιαίτερα, με ιδιαίτερα ερωτηματικά. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το συζητήσαμε αυτό και το συζητούμε ακόμα, δεν είναι καθόλου σαφές. Υπάρχει ένα μικρό έγγραφο εργασίας, αλλά ούτε αυτό είναι σαφές. Και βεβαίως, ξέρετε κύριε Επίτροπο, ότι την 1η Απριλίου υπήρξαν 16 χώρες οι οποίες σταμάτησαν ε, τα κοινωνικά ταμεία και άλλες τόσες τα περιφερειακά. Εντάξει, θα μπορούσαν να υπάρχουν προβλήματα για κάποιες χώρες, αλλά δεν είναι δυνατόν να έχουν πρόβλημα ρευστότητα όλες οι χώρες. Και τώρα σπρώχνουμε το σύνολο του προβλήματος το τελευταίο χρόνο, το 2013. Αυτό που λέει ο Επίτροπος είναι ότι εάν είναι πραγματικές αυτές οι πληρωμές θα πρέπει να αλλάξουμε τον προϋπολογισμό. Εγώ όμως λέω ότι απλώς ε, θα, θα σπρώξουμε τις οφειλές μέχρι το 2013 ε, και θα το βάλουμε μετά στο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το δεύτερο που θέλω να πω. Είπατε τις θέσεις σας. Λογικό είναι, είσαστε επίτροπος, λέτε τις θέσεις σας. Δεν σας ενδιαφέρει, λέτε, το θέμα των negotiation boxes Εμάς μας απασχολούν όμως ακόμα αυτά τα θέματα, τι σχετίζονται και με χρήματα, κάνουμε προτάσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί το σύνολο του οικοδομήματος και το πού πάνε τα χρήματα και αυτό παίζει ρόλο. Να σας πω όμως δύο πράγματα. Η εξάντε ερεσιμότητα δεν μετακινήστε από αυτό. Το ζήτημα είναι ε, θα πρέπει να συνδέσει αυτή την εξάντε με την απορροφητικότητα, με την απορρόφηση των, ε, ε, των πόρων στο Ταμείο Συνοχής, γιατί διαφορετικά δεν έχει καμία έννοια. Διαφορετικά θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Εγώ μπορώ να σας ε, δώσω στοιχεία και παραδείγματα για χώρες οι οποίες έχουν πολύ άσχημα μακροοικονομικά ε, στοιχεία, αλλά ήταν πάρα πολύ καλά όσον αφορά την απορρόφηση κονδυλίων ε, και ανάποδα, αντί, αντίστοιχα το ανάποδο. Όμως ξέρετε ότι ε, τα μακροοικονομικά προβλήματα κάποιων χωρών ενδεχομένως θα δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, την ήδη δυσχερή κατάσταση που αντιμετωπίζουν κάποιες περιφέρειες. Καλά θα ήταν όλα αυτά εάν δεν διανύαμε περίοδο κρίσης. Εάν δεν είχαμε διανύαμε περίοδο κρίσης, θα μπορούσαμε να θέσουμε ε, εκ των προτέρων και με μεγάλη έμφαση το θέμα της αιρεσιμότητας. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε αυτόν τον πολύ σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ε, στραθερότητας. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από πάνω κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω. Ε, τα αποθέματα αποδοτικότητας performance reserves. Εάν πρέπει να ε, εάν ε, κάνετε, βάλετε ένα 5% ε, στην αρχή ή στο μέσο της, των δημοσιονομικών προοπτικών, τότε οι χώρες ή οι περιφέρειες θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τον κίνδυνο αυτό και θα προτείνουν πιο εύκολα και όχι περίπλοκα προγράμματα. Γιατί τα περίπλοκα προγράμματα, τα οποία είναι και μακροχρόνια, ενδεχομένως διατρέχουν τον κίνδυνο στην ενδιάμεση αξιολόγηση να μην έχουν ολοκληρώσει κάποιο κομμάτι. Και τελικά δεν, τα προγράμματα τα οποία θα επιλεγούν δεν θα παράγουν ε, ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να απαντήσει σε αυτές τις τρεις παρεμβάσεις. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταρχάς, θα σας κάνουμε, θα σας διαθέσουμε μία ανακοίνωση για τα διαφορετικά ταμεία και τι πετύχαν πρόσφατα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας. Πάντα γίνεται διευκρίνηση ε, για τα θέματα αυτά. Πάντα ακούμε ότι δεν πρέπει να ακούμε τον όρο το unspent funds, ε, unused funds, γιατί όπως ξέρετε όλοι οι πόροι, όλα τα κονδύλια ε, χορηγούνται σε συγκεκριμένους προϋπολογισμούς. Δεν είναι χρήματα τα οποία πλέουν έτσι ελεύθερη, ελεύθερα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη διαχείριση των ε, προγραμμάτων, να περάσουν από τη μία από ένα κεφάλαιο στο άλλο κεφάλαιο, για παράδειγμα, του προϋπολογισμού, γιατί σε βλέπουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται όλο το κονδύλι, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις χρειάζονται επιπλέον χρήματα. Άρα τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω ότι έχουμε τροποποιήσει πιο, πολύ, πιο πολλά από 100 προγράμματα συνολικά. 17 δισεκατομμύρια συνολικής αξίας, 8 δισεκατομμύρια τους τελευταίους μήνες και λόγω χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία του Μπαρόσο που περιλαμβάνει και το ESF, γιατί εδώ μιλούσα μόνο για το EDF, θα υπάρχει ανακατανομή άλλων 5 έως 8 δισεκατομμυρίων που θα εστιαστούν στην καταπολέμηση της ενεργείας των νέων και της υποστήριξης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και πάλι, δεν έχουν γίνει συμφωνίες ε, με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο μπορεί να μας εμπιστεύεται σε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και η Επιτροπή αυτή αποτελεί τμήμα της διαπραγματευτικής ομάδας του Κοινοβουλίου έναντι του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, συγγνώμη. Δεν γνωρίζω επακριβώς τον τρόπο διαπραγμάτευσή σας, αλλά νομίζω ότι είναι γεγονός ότι είναι πλήρης ο ρόλος που διδραματίζει η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης στο ιστορικό του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις εταιρικές σχέσεις. Η ιδέα του Συμβουλίου είναι να το, να το αποκαλεί συμφωνίες. Ε, αλλά έτσι όπως κατανοούμε εμείς τις συμφωνίες αυτές στην ουσία έχουν ισχύ σύμβασης. Ε, έτσι όπως κατανοούμε την κατάσταση ε, είναι ότι η σύμβαση καλύπτει τα πάντα και όχι ορισμένα τμήματα και ορισμένα στοιχεία. Αυτό που δεν δεχόμαστε παραδείγματος χάρη είναι ότι κάποια στοιχεία της σύμβασης της εταιρικής σχέσης και του προσανατολισμού της εταιρικής σχέσης δεν θα ε, περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αυτή η αποστολή της ε, στρατηγικής ε, καλύπτει ήδη κάποιες απαιτήσεις. Ε, αυτό που κατανοούμε εμείς είναι ότι οι διαπραγματεύσεις και η αποδοχή του περιεχομένου της στρατηγικής ε, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην εταιρική σχέση. Όσον αφορά το θέμα των ΡΑΛ, υπάρχει εδώ μια παγίδα, ας πούμε, γιατί Εάν δεν έχουμε ε, αρκετό προϋπολογισμό, τότε ε, αναβάλουμε τις ε, πληρωμές και τότε φαίνεται να έχουμε αυξημένα ραλ. Πρέπει να, να είμαστε σαφείς και να είναι σαφές το τι κάνουμε απέναντι στα κράτη-μέλη. Οπωσδήποτε θα ζητήσουμε κάποια τροποποίηση του παρόντος προϋπολογισμού γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούμε στην κατάσταση στην οποία ε, περιγράψατε. Αυτό που θα ήθελα να πω σαφώς πάντως είναι το εξής, έστω και αν χρησιμοποιείται το επιχείρημα αυτό από κάποιες ε, χώρες μέλη, κυρίως από τους Υπουργούς ε, Οικονομικών, πρέπει να πω, λέω, ότι δεν υπάρχει ε, διαφοροποίηση ανάμεσα, στις, ε, ανάμεσα ε, στην αναβολή των πληρωμών και τα προβλήματα ρευστότητας από τη μία και το, το προσανατολισμό και τις αποφάσεις από την άλλη. Εάν υπάρχουν οποιασδήποτε καθυστερήσεις πληρωμών, αυτό οφείλεται σε ελλείψεις επιτόπου, που πούμε, και όχι όμως στην ροή του χρήματος. Επίσης, μετά από τα δύο τρίτα ας πούμε της ε, περίοδου ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει κάποια ενδιάμεση έτσι, αναθεώρηση που δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να είναι ακριβώς στη μέση της ε, ε, περίοδου και η performance ε, reserve θεωρητικώς ε, θα ε, μπορούσε να μειώσει την φιλοδοξία κάποιων χωρών ή κάποιων περιφερειών, αλλά γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε τα συμβόλαια εταιρική σχέσης, τα οποία καλύπτουν όλες τις διαπραγματεύσεις και που δεν μπορούν ας πούμε, να χρησιμοποιηθούν σαν πρόφαση από τις χώρες μέλη για να προτείνουν κάτι το οποίο θα είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξο από ό,τι θα όφιλε να είναι ε, είναι κατά την άποψή μας ε, ένα απαραίτητο κίνητρο και για τις χώρες ε, και για τις κυβερνήσεις δηλαδή και για τις περιφέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμα δύο συντονιστές. Αλφονσί, πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να σας στηρίξουμε σε αυτήν την ε, ε, σταθερότητα την οποία καταδεικνύεται έτσι ώστε το 14, στην περίοδο 14-20 ε, να είμαστε πολύ σαφείς όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής. Κατά την άποψή μας η πολιτική συνοχής έχει, αποδειξει, έχει αποδεικτεί ότι είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης και επομένως θα πρέπει να δοθούν στην Ευρώπη οι δυνατότητες να ε, ξεπεράσει την ε, κρίση, ε, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και σεβόμενη και τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές αρχές και να βασιστεί φυσικά και σε καινοτόμες πολιτικές όπως επανειλημμένα έχουμε πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ομάδα μας αλλά και πολλοί συνάδελφοι που είναι εδώ παρόντες εμείς υπερασπιζόμαστε την πολιτική συνοχή στα πλαίσια των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Η δράση σας ως ε, Επίτροπος ε, μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε πολλές ανταλλαγές απόψεων εδώ και το έγγραφο το οποίο μας υποβάλλεται ήδη εντάσσει ε, και περιέχει πολλά στοιχεία τα οποία έχουν προηγούμενα συζητηθεί εδώ ας πούμε το ζήτημα του νέου σχεδιασμού, των μεταβατικών περιοχών, ε, άλλα καινοτόμα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην ε, πολύ ενδιαφέρουσα κατά την άποψή μας ε, πρόταση θα ήθελα τώρα να αναφερθώ και στα σημεία τα οποία δεν μας αρέσουν πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ε, θα μιλήσω σαν εκπρόσωπος νησιωτικής ε, περιοχής. Έχω μιλήσει και με άλλους νησιώτες ε, βουλευτές και έχουμε την εντύπωση ότι δεν μας έχει καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει καταλάβει τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουμε. Στρεφόμαστε λοιπόν προς εσάς κύριε Επίτροπε και ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις μας. Δεύτερον, Υπάρχει το πρόβλημα της ε, μακροαιρεσιμότητας, ε, το οποίο έθιξαν κι άλλοι ε, συνάδελφοι. Ξέρουμε ότι αυτή η πρόταση προωθείται από κάποιες χώρες, αλλά επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι κατά την άποψή μας δεν είναι λογική και δεν είναι και συνεπής. Δηλαδή δεν δίνει το αποτέλεσμα το οποίο υποτίθεται ότι θέλει να δώσει. Ε, και αντιθέτως ε, θα επιδεινώσει σε μερικές περιπτώσεις την κατάσταση σε ορισμένε χώρες. Έχουμε σήμερα ε, ένα 38 παράδειγμα, ένα φωναχτό παράδειγμα με την Ελλάδα, αλλά μην ξεχνάτε ότι μέχρι το 2020 πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι πολλές χώρες ακολουθούν το παράδειγμα της Ελλάδας και επομένως δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν πρέπει να βάλουμε και περισσότερα εμπόδια στην ορθή λειτουργία του συστήματος. Κάνω λοιπόν έκκληση τη στιγμή που η ε, πολιτικοί συσχετισμοί και οι πολιτικές ισορροπίες φαίνεται να αλλάζουν λίγο στην Ευρώπη. Ε, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουν και κάποιες ε, άλλες αρχές. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Αλφόνση και Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι ιδιαιτέρως χαίρομαι διαπιστώνοντας ε, την προσωπική σας ε, δέσμευση στην προώθηση της αστικής διάστασης, γιατί τα χρήματα τα οποία δίδονται στην αστική διάσταση και στις πόλεις και στις γενικότερες εδαφικές ε, μονάδες ε, οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία τα οποία χρήζουν από Πρώτα απ' όλα, αυτό το 5% για τις πόλεις, ε, η ερώτησή μου είναι ποια είναι τα σχέδια, τα project τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο 5%. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. δεύτερη ερώτηση αφορά την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε την κατηγορία αυτή έτσι ώστε να περιληφθούν και κάποιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τουλάχιστον να μην ε, αποκλειστεί κάποια εταιρεία, έστω και αν αυτή είναι μια μεγάλη ε, επιχείρηση ας πούμε. Ε, και επίσης μην ξεχνάτε ότι οι μεγάλες ε, εταιρείες πολύ συχνά έχουν υπεργολάβους ε, και προμηθευτές μικρότερες εταιρείες. Θα πρέπει να δούμε ποιους θέλουμε να στηρίξουμε και ποια θα είναι η καλύτερη προσέγγιση έτσι ώστε να επιτύχουμε τους στόχους συνοχής και, τη στρατηγική, και τους στόχους της στρατηγικής 2020 όσον αφορά την αηφόρο στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε μονάχα στην άμεση στήριξη. Θα πρέπει να προωθήσουμε γενικότερα την οικονομία, ε, έτσι ώστε να βελτιωθούν καλύτερα όλοι όσοι ε, βρίσκονται στην αλυσίδα ε, της μεταποίησης, του εμπορίου κτλ. Θέλουμε αστική ανάπτυξη, αλλά θέλουμε και ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα ήθελα να μου πείτε και την άποψή σας ε, για το ε, CEF. Τελευταίο σχόλιο. Η διαπραγματευτική μας ε, θέση είναι πιο δύσκολη διότι οι προτάσεις αυτές θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί από την Κομισιόν στα τέλη του προηγούμενου χρόνου, αλλά τελικά υπευλήθησαν αργότερα, πολύ αργότερα, τον Μάρτιο. Η κατάσταση είναι, είναι δυσκολότερη και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Με μονομένες παρεμβάσεις τώρα, αλλά να σας ζητήσω να μην υπερβείτε ο καθένας σας τα τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σρέντερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να επανέλθω στην ε, τελευταία, στο τελευταίο τμήμα της εισήγησή σας, κύριε Επιτροπέ, όπου είπατε ότι απευθύνεται μια μεγάλη έκκληση εδώ στο Κοινοβούλιο. Ναι, θέλουμε μια αυστηρή πολιτική συνοχή με βάση συγκεκριμένους, συγκεκριμένα θέματα. Αυτό θέλουμε και εμείς, αλλά κοιτώντας τον κανονισμό βλέπουμε ότι κάποια μέσα είναι ίσω υπερβολικά αυστηρά σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό τους στου θεματικού στόχους και δεν έχουν λάβει υπόψη το γεγονός ότι και αλλιώς μπορούν να εφαρμοστούν οι θεματικοί αυτοί οι στόχοι και τα πράγματα δυσκολεύουν με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν είναι και καλύτερη η ε, πρόταση του Συμβουλίου, αν και εμείς συμφωνούμε ως πράσινοι, γιατί όπως είπε ο συνάδελφος Φλάζακ, ε, ε, θέλουμε μια ενεπιμενή προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ε, ότι ως Επίτροπος προς αυτή την κατεύθυνση κινείστε. Ότι λέμε δηλαδή ότι εντάξει σε έναν άξονα προτεραιότητας ε, μπορούμε να έχουμε μια ενοποίηση χωρίς ε, να πρέπει να ζητάμε χρήματα από κάθε υπηρεσία για οποιαδήποτε ενοποιημένη προσέγγιση. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να ξανασκεφτείτε λίγο την προσέγγιση σας και ανυπομονώ να ακούσω ποια είναι η αντίδρασή σας. Äh, σε ό,τι αφορά την μακροαρεσιμότητα. Νομίζω ότι σε πολλές περιστάσεις έχουμε ανταλλάξει απόψη το θέμα αυτό και η τρέχουσα κατάσταση νομίζω καταδεικνύει πόσο απαραίτητο είναι το στοιχείο αυτό να εξακολουθήσει να θεωρείται ενδεχόμενο μέσο. Γιατί διασφαλίζει ότι ουσιαστικά περιλαμβάνονται όλα τα κράτη-μέλη. Οι μηχανισμοί κυρώσεων ισχύουν μόνο για, τα, για τις του ευρώ. Και αυτό δεν θα ήταν σωστό από κάποια άποψη σε ό,τι αφορά τώρα τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Βρισκόμαστε σε φάση συζήτησης, αλλά θα ήθελα να υποδείξω ότι ο τωρινός και ο μελλοντικός κανονισμός δίνουν πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης προκειμένου να ανταποκριθούμε στις δημορφίες αυτές. Αλλά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις και είμαστε στη διάθεσή σας. Για τον συνάδελφο Βλάσακ, να σας ευχαριστήσω για την ε, ε, υπόδειξη στην αστική διάσταση. Αλλά θα ήθελα να σας πω ανοιχτά ότι στις διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο ιδιαίτερα η αστική διάσταση και η ειδική ε, χρηματοοικονομική διαμόρφωση δεν οδήγησαν στο να δημιουργηθεί μία αλλαγή τέτοια. Ήταν κριτική η στάση. Και στο σημείο αυτό θεωρούν πολύ ότι υπάρχει δυναμικό και δυνατότητα εξοικονόμησης ε, χρημάτων. Θα ήθελα να σας υποστηρίξω και να σας ενθαρρύνω σε ό,τι αφορά την άποψη σας αυτής για το 5%. Είναι κατώτατο το όριο αυτό και σκοπό έχει να χρηματοδοτήσει ενοποιημένες περιφερειακές πρωτοβουλίες, κυρίως όταν ε, εγγυάται ότι η διαχείριση θα είναι κυρίως στα χέρια του κράτους μέλους. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Μου ζητήσατε ένα παράδειγμα για την ε, αναζωγόνηση μιας ε, παρεκμασμένης, για παράδειγμα, πόλης, ενός παρικμασμένου τμήματος μιας πόλης. Υπάρχουν διάφορα μέσα τα, μπορεί τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν. Μιλάμε για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ε, υγείας. Μπορεί να απασχολεί, να αφορά μάλλον ε, δυνατότητες απασχόλησης σε κάποιο τμήμα. Και κατά πάσα πιθανότητα τη βελτίωση του οικιστικού επίπεδου σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ε, ενεργειακό ζήτημα ε, ή για παράδειγμα ζητήματα μεταφοράς. Το θέμα λοιπόν είναι ένα τμήμα μιας πόλης το οποίο έχει ε, παρακμάσει να τονωθεί. Αυτά μπορούν να πετύχουν μόνο αν χρησιμοποιηθούν δέσμες μέτρων από διάφορους τομείς. Και αυτό με οδηγεί στο δεύτερο θέμα σας, ε, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό, θεωρώ, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την πρότασή μα, ήδη σήμερα οι μεγάλες επιχειρήσει όταν δραστηριοποιούνται ε, σε θέματα ενέργειας και έρευνας μπορούν να λάβουν υποστήριξη. Αυτό θα παραμείνει γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας. Όταν όμως πρόκειται καθαρά για θέματα επένδυσης επιχειρησιακών μέσων κτλ. Θεωρούμε από την εμπειρία μας ότι δεν είναι απαραίτητο να ενισχυθούν. Για κάποιους τομείς, λοιπόν, η πρότασή μας περιλαμβάνει δυνατότητα ενίσχυσης και στα πλαίσια μεγάλων επιχειρήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου, προσπαθήσαμε μεταξύ άλλων και μεταξύ μέσω του στρατηγικού πλαισίου, να κάνουμε διευκρινήσεις για το τι πρέπει να κάνει ποιος και πού. Και ναι, υπήρχε μια καθυστέρηση στην παρουσίαση του κοινού αυτού στρατηγικού πλαισίου. Αυτό οφείλεται στο ότι ήταν η πρώτη φορά και σε κάποιες περιπτώσεις η φιλοδοξία είναι λίγο πιο ε, μεγάλη σε ό,τι αφορά το χρονικό περιθώριο. Αλλά βασικά αυτό που μας απασχολούσε στις υπηρεσίες της Επιτροπής είναι να μην ε, προτιμήσουμε την ταχύτητα από την ποιότητα. Να προτιμήσουμε την ποιότητα ή βάρος ίσως της ταχύτητας. Ελπίζω στο κοινό αυτό στρατηγικό πλαίσιο να, μάλλον το κοινό στρατηγικό πλαίσιο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Για την κυρία Σουρέντερ τώρα. Εμείς πάντα είμαστε ανοικτοί να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι το εξή ότι αν ε, επιδείξουμε υπερβολική χαλαρότητα και γενεοδορία, και αυτό βλέπω στις συζητήσεις σήμερα, αν προσθέσουμε υπό το πνεύμα της ευελιξίας ε, όλα τα δυνατά στοιχεία, τελικά θα καταλήξουμε σε μία αντίφαση. Στόχος μου λοιπόν πάντα είναι να έχουμε την επικέντρωση, να υπάρχει κάποια ευελιξία σε ό,τι αφορά τους τομείς κατανομής για τις βασικές προτεραιότητες, για παράδειγμα το θέμα των βιώσιμων αστικών μεταφορών, ασφαλώς θα πρέπει και αυτό να μπορεί να συμπεριληφθεί ως μέτρο ε, ενεργειακής αποδοτικότητας, προκειμένου να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό. Αλλά αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς, νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί και μέσω των multi και των ε, διευρυμένων δυνατοτήτων στα multi-funds, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιβαρύνεται και διακυβεύεται η συνολική στοχοθεσία. you very much. Jan Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάν Όλμπριχτ. Ένα πολιτικό και τρία τεχνικά σχόλια. Πρώτα απ' όλα με επιτρέπετε το πολιτικό σχόλιο και ερώτημα. Τι σχέση, έχει υπάρχει μεταξύ των φίλων της συνοχής και των φίλων της ε, καλής ε, δαπάνης, αν μπορώ να το πω έτσι, της ορθολογικής δαπάνης. Πώς ε, διαγράφεται η κατάσταση. Ποια είναι η άποψη της Κομισιόν, γιατί κατά τη δική μας άποψη δεν είναι σε παράθεση οι δύο πλευρές. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο λιγμού. Εσείς τι έχετε να μας πείτε από αυτού. Δεύτερο, ένα τεχνικό ζήτημα. Σε ποιο βαθμό η έλλειψη συμφωνίας ε, στο, στις διαπραγματεύσεις για τον δημοσιονομικό κανονισμό επηρεάζει και το νομοθετικό έργο. Το γεγονός ότι το άρθρο 56 ακόμη δεν έχει τύχει συμφωνία, σε επηρεάζει κατά την άποψή σας την νομοθετική διαδικασία και την όλη δυναμική. Αν τώρα πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στον προϋπολογισμό και οι περικοπές αυτές προφανώς θα επηρεάσουν και την πολιτική συνοχής. Το ερώτημά μου, και είναι ένα ερώτημα που έχω επαναλάβει πολλές φορές, πώς θα γίνει η περικοπή αυτή. Μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε από το Connecting Europe. Θα μπορούσαμε να έχουμε τεράστιες εξοικονομήσεις πόρων. Εντάξει, να εξοικονομήσουμε δέκα δις, όχι, αυτό είναι αδύνατο, αλλά θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε πολύ περισσότερα κονδύλια στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών. Υπάρχουν ε, παρανοήσεις για το από πού μπορούν να βρεθούν, από πού μπορούν να γίνουν οικονομίες. Υπάρχουν βέβαια και πολιτικοί στόχοι της Κομισιόν και το καταλαβαίνω. Εγώ πάντως θα καταθέσω σχετικές τροπολογίες για την πλήρη διαγραφή του Connecting Europe από τον κανονισμό. Τελευταία μου παρατήρηση. έχει να κάνει με τη θέση σας, τη δική σας θέση κύριε Επίτροπε. Αυτό που εμείς αντιλαμβανόμεθα ως θεματική συγκέντρωση, επικέντρωση και αυτό το οποίο από την άλλη ε, εννοούμε ως ευελιξία, εκεί υπάρχει κάποια αντίφαση, κάποια προβλήματα υπάρχουν. Πολλές φορές έχει πει ο πρόεδρος Μπαρόζο ότι σε καιρό κρίσης αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια γρήγορη αλλαγή, μια ταχεία μεταβολή σε ό,τι αφορά δηλαδή τον επαναπρογραμματισμό. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι ευέλικτα μέσα και εργαλεία. Αν πρέπει να είναι αυτά τα μέσα λοιπόν ευέλικτα, δεν μπορεί να τα περιχαρακώσουμε και να τα καταστήσουμε άκαμπτα, γιατί αυτό είναι αντιφατικό εξορισμού. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι η θεματική συγκέντρωση ως μια δέσμη στόχων απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Στη δική μου έκθεση προτείνω οι μεταφορές να μεταφερθούν στην θεματική συγκέντρωση με το εξής σκεπτικό. Πρέπει να περιορίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και που είναι πολύ σημαντικός εδώ ο τομέας των μεταφορών. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, και αν ο στόχο αυτό επίση είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να δούμε αυτέ τι θέσει δημιουργούνται μόνο από μικρομεσαίε επιχειρήσει ή μπορούν να τι δημιουργήσουν και κάποιε μεγάλε επιχειρήσει. Πού επικεντρώνουμε την προσοχή μα περισσότερο, στη δημιουργία θέσεων εργασία ή στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρέπει να επιλέξουμε την προσέγγιση. Εντάξει, ναι στην ε, θεματική συγκέντρωση, επικέντρωση, συμφωνούμε. Αλλά Εάν θέλουμε να έχουμε έναν πιο ευέλικτο επαναπρογραμματισμό, οι δικαιούχοι και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια, μεγαλύτερη ελευθερία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίφαση σε αυτό. Σας ε, ανέφερα λοιπόν τα ερωτήματά μου. Περιμένω κάποιες απαντήσεις. Κύριος Μποστινάρου, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το οποίο θα σας πω ευθύ αμέσω ευθυγραμμίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα όσα προείπε ο αγαπητός συνάδελφος Όλμπριχτ. Ναι, μεν ανήκουμε σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες, αλλά βλέπουμε ότι κάπου μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ καλά γνωρίζουμε ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν δύο ε, κατηγορίε. Οι φίλοι τη πολιτική συνοχή και οι φίλοι των πιο ορθολογικών δαπάνων, τη καλύτερη δαπάνη. Εμεί όμω έχουμε καταφέρει στην Επιτροπή μα να συγχωνεύσουμε αυτέ τι δύο ομάδε και ουσιαστικά μιλούμε την ίδια γλώσσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αγωνιζόμαστε δηλαδή για να υπάρχει μεγάλη στήριξη στην πολιτική συνοχή, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε απτά ωφέλη, απτά αποτελέσματα, τα οποία είναι αισθητά σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων. Εκείνο από αυτό λοιπόν, θέλω να σας πω τα εξής. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει αυτόν τον ουδέτερο ρόλο μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Είναι ξεκάθαρο είναι ηλίου φαϊνότερο για εμένα τουλάχιστον ότι όσοι αγωνίζονται υπέρ της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να είναι όχι μόνο εταίροι αλλά θα πρέπει και να μιλούν την ίδια γλώσσα για να μπορέσουν τελικά να πείσουν και το Συμβούλιο ότι γιατί το πάτε κι εσείς. Είναι σημαντικό για την ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων απασχόλησης πώς μπορούμε να περάσουμε πλέον από μέτρα λιτότητας σε αναπτυξιακά μέτρα. Και βέβαια έτσι θα σώσουμε στο τέλος και την Ευρώπη, γιατί η λιτότητα μπορεί να σκοτώσει το κοινό μας αυτό ε, σχέδιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή σχέση και συνεργασία που είχαμε προσωπικά μαζί σας αλλά και με τη ΓΔ κατά τη σύνταξη των εκθέσεών μας και στη διάρκεια των συζητήσεών μας. Είμαι πεπισμένος ότι θα συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία. Και τώρα, για να ολοκληρώσω, κύριε Επίτροπε, και πάλι συμφωνώντας με τα σχόλια του συναδέλφου Όλμπριχτ, πώς αξιολογείται σήμερα την κατάσταση με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, διότι έχουμε από τη μια πλευρά άτομα που στεναρά αντιτίθενται σε αυτό το πλαίσιο στο Συμβουλό, σημαντικα σημαντικά κράτη-μέλη και αρκετά πολλά, και από την άλλη πλευρά, εντό Ευρωκοινοβουλίου υπάρχει μια αντίσταση, αλλά υπάρχουν και άλλοι μεταξύ αυτών και εγώ, που θέλουμε να έχει ωφέλη και αποτελέσματα το στρατηγικό πλαίσιο, αλλά να συμβαδίζει ταυτόχρονα με και την ε, φιλοσοφία μας περί συνοχής. Και να μην επικρατεί μόνο το TNT για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ίσως να έχετε υπόψη σας ότι ορισμένοι από εμάς επανειλημμένως επιχειρήσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΜΟΥΒ. Ζητούμε από εσάς και από τον Επίτροπο Κάλλας να μιλήσετε την ίδια γλώσσα για αυτά τα θέματα. Μπορεί να γνωρίζετε όμως ότι ο Επίτροπος Κάλλας τις τελευταίες ημέρες είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά των 10 η μεταφορά δεν πρόκειται να περάσει σε καμία περίπτωση το ανώτατο όριο. Αυτό είναι απίστευτο, είναι αδύνατο. Ή θα μεταφερθούν οι πόροι από το Ταμείο Συνοχής, γιατί ε, η δική μου έκθεση αυτό ακριβώς αφορά, ή θα πέσουν μου αυτο ακριβως αφορα η θα πεσουν απο τον ουρανό αυτά τα χρήματα. Δεν νομίζω θα μας, ε, θα μας πέσουν από τον ουρανό λεφτά, σήμερα τουλάχιστον. Πού θα βρεθούν τα λεφτά, τα λεφτά λοιπόν, πρώτον και δεύτερον, θα υπάρχουν όρια να μεταφερθούν. Γιατί ε, σίγουρα πρέπει να εξομαλύνουμε τις εντάσεις και να ε, μειώσουμε κάπως ε, την ε, αντιπαράθεση. Πώς εξελογείται λοιπόν την κατάσταση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Νούνιο Τεσέρα, τελευταίος ομιλητής. Είχατε αποκοιμηθεί, σας ξύπνησα. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν με είχε πάρει ο ύπνο σε καμία περίπτωση, κυρία Πρόεδρε. Ε, λίγο είχε έτσι γύρει το κεφάλι. Τέλο πάντων, λοιπόν, τρία ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες ημέρες, 2 ή 4 Ιουλίου, θα ε, οργανώσει ένα φόρουμ για τις ε, ακρος απόμακρες περιοχές. Ε, υπάρχει συντονισμός με κάποιες εργασίες που γίνονται. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου πρόσφατα ενέκρινε μία έκθεση ακριβώς για το ίδιο θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω εκ ότι εγώ διαφωνώ. Η Κομισιόν δεν απέδωσε την δέουσα προσοχή Εμείς είμαστε στο Στρασβούργο εκείνη την εβδομάδα. Δεν θα μπορέσουμε να λάβουμε μέρος. Θα έπρεπε να φροντίσετε να μπορεί να είναι παρόν και το Κοινοβούλιο. Δεν μας ε, βολεύουν αυτές οι ημερομηνίε. Πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία. Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να γίνουν έτσι τα πράγματα. Έρχομαι τώρα σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Για το ΦΕΝΤΕΡ, λοιπόν, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ξέρετε, υπάρχει για τις ε, άκρος απόκεντρες ε, περιφέρειες ένα συγκεκριμένο κονδύλι και υπάρχουν ε, και κάποιες περικοπές για τις μεσημερινές περιοχές. Για το 2013 προβλέπονται ακόμα μεγαλύτερες περικοπές. Πώς τα δικαιολογείτε εσείς όλα αυτά. για την ανταγωνιστικότητα, για την απασχόληση. Υπάρχουν περιοχές πολύ ανεπτυγμένες ε, με πολύ μεγάλο ΑΕΠ. Έχουμε ένα 3% σε 55 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει περικοπή μόνο 3% για αυτές τις περιφέρειες, ενώ για άλλες που προβλέπεται μείωση κατά 47%. Επόμενο ερώτημα. Υπάρχουν κάποιες ε, χαμηλές, χαμηλά ποσοστά ε, χρησιμοποίησης. Αυτό είναι ο λόγος. Γιατί τότε το ποσοστό χρηματοδότηση παραμένει στο 50% και δεν εναρμονίζεται το 50% με το 85% της συγχρηματοδότησης που προβλέπεται για τον κανονισμό ε, του ΕΤΠΑ και για τις άκρως απόκεντρες ε, περιφέρειας. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Ε, δεν καταλαβαίνω, θα ήθελα λοιπόν να μου το εξηγήσετε. Τρίτη και τελευταία ερώτηση. Παρακολούθησα με πάρα πολύ ενδιαφέρον την παρέμβασή σας και είπατε ότι αν ευελιξία σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με τα κονδύλια, δεν θα πετύχουμε ποτέ το στόχο της βιωσιμότητας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτή σας τη δήλωση. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι σε ό,τι αφορά αυτά τα ειδικά κονδύλια, αυτή την ειδική πρικοδότηση, υπάρχει υποχρέωση το 50% αυτού του ποσού να αποδοθεί στην θεματική συγκέντρωση. Και αυτό περιλαμβάνεται στο γενικό κανονισμό για το Ταμείο. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Γιατί για τι άκρω απόκεντρε περιφέρειε υπάρχει αυτή η υποχρέωση το 5% τη ειδική προκοδόκηση να μπει σε στόχου θεματική συγκέντρωση, αλλά για τι βόρειε αεροκατοικημένε περιοχέ δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση θεματική συγκέντρωση. Εδώ λοιπόν χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά και δεν το καταλαβαίνω. Θα ήθελα λοιπόν να μου το εξηγήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Επίτροπο έχει το λόγο. <clears throat> Ε, για τον κύριο Όλμπριχτ. Στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου μίλησα για το better spending και ζήτησα ως σύμβολο οικοδόμησης γεφυρών να γίνει αυτό, γιατί δεν βλέπω ότι υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις Ελπίζω η ομάδα Better Spending να προσεγγίσει τους Friends of Cohesion και να κατανοήσουν ότι η καλύτερη δαπάνη των κονδυλίων μπορεί να έχει αποτελέσματα ίσως με διαφορετική στοχοθέτηση, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντιφάσεις ουσιαστικά. Αυτή είναι η θέση μου λοιπόν και την ε, αναφέρω σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς κανονισμούς τώρα. Όντως, υπάρχει ο κίνδυνος, αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, να πληχθούμε στη φάση της οριστικοποίησης. Ελπίζω αυτό το άρθρο 56, το περίφημο, να καταλήξει σε συμφωνία, προκειμένου να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την θεματική κατάστασης Αν η ιδέα ήταν για ένα project να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά κονδύλια, έχουμε τις επιφυλάξεις μας, αλλά δεν είναι επί της αρχής τόσο πολύ. Ναι, μα να μιλάω μόνος μου αν θέλετε. κάποια γλωσσικά καθεστώτα είναι λίγο πιο ηχηρά φαίνεται. Για λόγους λοιπόν διαχείρισης αντιμετωπίζουμε δυσκολίες να εφαρμόσουμε διάφορα κονδύλια σε ένα project, σε ένα έργο. Αλλά υπάρχει αυτή η προσέγγιση multi-funds, η θεματική επικέντρωση. Αυτό που με ανησυχεί είναι το εξής. να προωθηθούν ε, βασικές ε, υπηρεσίες ε, σε περιφέρειες, για παράδειγμα σε θέματα μεταφοράς. Υπάρχουν κάποια όρια για την ενίσχυση. Πολλές περιφέρειες μπορώ να σας αναφέρω στην Ευρώπη που λαμβάνουν χαμηλά ποσά και η επένδυση για παράδειγμα σε ένα δρόμο θα σήμαινε ότι θα εξαντλούνταν όλα τα κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν οι προτάσεις μας ε, έχουν να κάνουν με τον περιορισμό. Αυτό είναι πρακτικό το θέμα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων έναντι της υποστήριξης των ε, μεγάλων επιχειρήσεων. Να σας πω ως πρώην διευθυντής Μεγάλου Ομίλου ότι όταν αν λάβαμε όταν λάβαμε τις βασικές αποφάσεις μας, ε, τρία θέματα μας απασχόλησαν. Κράτος δικαίου. Υπάρχει μία τάση να αλλάζουν αναδρομικά νομοθεσίας. Δεύτερον, νομοθετικό ε, φορολογικό πλαίσιο. Και τρίτον, διαθεσιμότητα ε, εξειδικευμένου προσωπικού. Γιατί δεν μπορώ όταν ανοίγω κάπου ένα εργοστάσιο, μια ταση να αλλαζουν αναδρομικα νομοθεσιας δευτερον νομοθετικο φορολογικο πλαισιο και τριτον διαθεσιμοτητα ε προσωπικου γιατι δεν μπορω οταν ανοιγω καπου ενα εργοστασιο μια εταιρεια να φέρναμε το αεροπλάνο τους εξειδικευμένους ε, συνεργάτες. Αυτά ήταν τα τρία θέματα που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα. Το θέμα της ενίσχυσης είναι, όπως λέμε, nice to have, καλό για τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, αλλά καθοριστική είναι, καθοριστικές είναι αυτές οι τρεις παράμετροι. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο που έχουμε περιορισμένα μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκεί που πραγματικά είναι απαραίτητα για να ρυθμίσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και νομίζω ότι στο σημείο αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους είναι ωφέλιμη. Αλλά όταν μιλάμε για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, για παράδειγμα, νομίζω ότι ως κοινωνία έχουμε συμφέρον και θα πρέπει να τα προσφέρουμε αυτά στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ε, δουλεύουμε με, με τα revolving funds. Αν θέλουμε να, υπάρχει αποτελέσματα, να υπάρχουν αποτελέσματα και από πλευρά των επιχειρήσεων. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να παρέχουμε γιατί και εμάς μας συμφέρει. σε ό,τι αφορά το Connecting Europe Facility. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα αυτό και πρέπει να γίνουν και άλλες συνδέσεις προκειμένου να υπάρχει όντως αυτό το μέσο ως facility. Νομίζω ότι η πρόταση που έχουμε στη διάθεσή μας είναι σαφής. 10 δις, όπως προτάθηκε από τον προπολογισμό, 10 δις από τα ταμεία συνοχής με κανέναν άλλον περιορισμό και αυτό συζητιέται φυσικά και αυτή θα πρέπει να είναι η συζήτηση για τις ε, ε, αποκεντρεμένες περιοχές. Ζητώ συγγνώμη για την ημερομηνία αυτή, αλλά η συνεδρίαση γίνεται Δευτέρα πρωί ε, στις Βρυξέλλες και μετά έχουμε Στρασβούργο το μεσημέρι συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Ίσως ε, υπάρχει κάποια δυνατότητα να συμμετάσχει κανείς και στις δύο συνεδριάσεις. Εγώ έχω μία θέση στο αυτοκίνητό μου να προσφέρω, γιατί σίγουρα θα πάω μετά στο Στρασβούργο. Σε ό,τι αφορά τη μείωση Ναι, κάναμε μειώσει στα special allocations, αλλά κάναμε και μία πρόταση σαφούς αύξηση των μέσων σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό συνεργασία, το οποίο είχαν ζητήσει πολλέ αποκεντρωμένε ε, ε, περιοχές. Άρα, αν τα συνυπολογίσουμε αυτά, η μείωση και η περικοπή είναι πολύ πιο περιορισμένη. Το 50% που είχαμε προτείνει στα special allocations έχει να κάνει καταρχάς με τη διεύρυνση της οικονομικής ε, ε, δραστηριότητας της αποκεντρωμένης περιοχής και λέω ξεκάθαρα ότι στόχος μου είναι οι αποκεντρωμένες περιοχές οικονομικά να γίνουν βιώσιμες και αυτόνομες. Αυτή είναι η στοχοθεσία μας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε πολλές τέτοιες περιοχές μόνο όταν το φάσμα των δραστηριοτήτων διευρυνθεί σε ό,τι αφορά τις οικονομικές δραστηριότητες και απαλλαγούν από οικονομικές ε, μονολυθικές δραστηριότητες, αν υπάρξει ένα εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων. Γι' αυτό λοιπόν τα ήπια μέσα του 50% των κονδυλίων προτείνεται λοιπόν να χρησιμοποιηθούν έτσι. Και για θέματα συγχρηματοδότησης και ποσοστούς συγχρηματοδότησης θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τσέλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι μιλάνε για ανάπτυξη και λες και ένα φάντασμα να περνάει στην Ευρώπη ότι χρησιμοποιούμε την ε, ανάπτυξη για να καταπολεμήσουμε την κρίση. Αλλά πού θα βγει αυτή η ανάπτυξη, κανείς δεν το αναφέρει αυτό και με, ποιους, ε, με ποιες μεθόδους. Και κράτη-μέλη τα οποία πριν από ένα χρόνο ούτε ήξεραν τι είναι η περιφερειακή πολιτική. Τώρα μιλάνε για περιφερειακή πολιτική και λένε ότι θα δημιουργήσουν ανάπτυξη. Υποθέτω ότι εννοούν ότι ανάπτυξη εννοούν την αύξηση του ε, ΑΕΠ της ε, χώρας τους. Γιατί η μείωση του ΑΕΠ προκαλείται από την ε, κατάρρευση του τραπεζικού τομέα, από την κατάρρευση ενός σημαντικού τμήματος του τομέα των ακινήτων στην Ισπανία, της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γαλλία. Μείωση των ε, επιδοτήσεων ε, ηλιακών ε, εγκαταστάσεων στη Γερμανία και αυτό οδηγεί σε κατάρρευση πολλέ πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα νέα στα νέα ομοσπονδιακά κρατήρια και όλα αυτά θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με τα αντιστατικά ταμεία. Και εκ παραλίλου ανακαλύψαμε και αυτό το υποτιμάμε ότι έχουμε 83 δισεκατομμύρια τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ακόμα και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Απασχόλησης ε, μας είπαν ότι, κοιτάξτε, έχουμε 83 δισεκατομμύρια ε, μη απορροφημένα κονδύλια περιφερειακής ανάπτυξης. Θα τα χρησιμοποιήσουμε για προγράμματα ε, απασχόλησης, κατάρτισης των νέων κτλ. Όποιος έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά και ξέρει τι σημαίνουν τα προγράμματα κατάρτισης για τους νέους, γνωρίζει πόσοι φορείς θα πρέπει να συμμετάσχουν και τι δαπάνη χρειάζεται. Και ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε αυτά τα χρήματα από την τσέπη μας ε, έτσι γρήγορα. Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν με τα αυτά μέσα. Σωστά είπατε και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε ότι έχουν οριστεί για την παρούσα προγραμματική περίοδο. Δεν υπάρχει ευελιξία εκτός και αν τα κράτη-μέλη, αν οι περιφέρειες που έχουν τη δυνατότητα και διαθέτουν τα κονδύλια αυτά συμφωνήσουν και θα πρέπει να συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια αυτά για άλλες δαπάνες. Τώρα σε ό,τι αφορά τη νέα προγραμματική περίοδο και τι εννοούμε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία συνοχή ε, για ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχει μια πιο κεντρική διαχείριση, δηλαδή τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά στους οικονομικούς τομείς εκείνους όπου θεωρούν ότι μπορούν να δώσουν οικονομικά κίνητρα. Αυτό τι θα σήμαινε όμως ότι η πολιτική συνοχή θα εγκατέλειπε την περιφερειακή διάστασή της αν θέλετε. Και αυτό τι θα σήμαινε επίσης και για τον τρόπο διαχείρισης ε, και τον τρόπο αντιμετώπισης της πολιτικής ε, συνοχής υπάρχει ο κανονισμός, καταρχάς τα λειτουργικά προγράμματα σε επίπεδο κρατών μελών, όπου υπάρχει και ομόσπονδο, ομοσπονδιακό κράτος, υπάρχουν και τα προγράμματα σε επίπεδο ομόσπονδων κρατηδίων και στην Αυστρία και στη Γερμανία υπάρχουν ε, τομεακά προγράμματα τα οποία επιβεβαιώνονται και αποτελούν την ε, βάση για τα επόμενα 7 χρόνια ή για τα εν συν δύο χρόνια. Και αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις κρίσης που έχουν τις αιτίες τους αλλά δεν προβλέπονται πάντα. Είναι απρόβλεπτοι παράγοντες. Αν θέλουμε να έχουμε δυνατότητα αντίδραση σε τέτοιες κρίσεις, αν θέλουμε να υπάρχει αυτή η εγγύηση των ρηστατικών ε, και ταμείων και ταμείων συνοχή, αν θέλουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση ταμείων κρίσης. Πώς το έχουμε φανταστεί, δεν βλέπουν να έχουμε τη δυνατότητα στην παρούσα φάση να παρέμβουμε οικονομικά. Τι θέλουμε, θέλουμε στο μέλλον ε, ταμεία παρέμβασης ε, ή θέλουμε ένα ταμείο καθοδήγηση στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου του Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, τι χαρακτήρα θέλουμε να έχουν αυτά τα ταμεία, να ενισχύσουν όπω όπως έκαναν ως τώρα τις περιφέρειες προκειμένου να μην χάσουν τα δυνατά του σημεία. Νομίζω ότι πρόκειται για μια συζήτηση επί της αρχής, η οποία θα πρέπει να γίνει τώρα. Ιδάλλως, το συζήτησα και με τον συνάδελφο Βίνκλερ, στην ε, Ανατολική Γερμανία, ξέρετε, όλοι μιλούσαν για την εκπλήρωση των βασικών καθηκόντων που ήταν ε, η εκπλήρωση της ε, κοινωνικής πολιτικής. Αυτό δυστυχώς δεν πέτυχε τότε, ξέρετε. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Όσοι είναι στον κατάλογο θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σύντομοι, γιατί μεγαλώνει ο κατάλογος των ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, για να μπορούν να αναπτυχθούν ορισμένες περιφέρειες πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στις υποδομές. Κάποιες άλλες περιφέρειες πρέπει να επενδύσουν σε πιο σοφιστική, αν μπορώ να τα πω, έργα. Δεν θέλω να σας δώσω ένα Παράδειγμα, είμαι πολικός μηχανικός. Αν ετοιμάσουμε ένα έργο οδικών υποδομών, οδοπία, πρέπει να το προετοιμάσεις, μετά να περάσει από τη διαδικασία του διαγωνισμού. Χρειάζεται καιρός. Στο μεταξύ, κάπου σε αυτό το δρόμο, ας πούμε, γίνεται μία ε, ζημιά. Δεν λειτουργεί καλά ε, και αν κάποιος παρεκκλίνει από το έργο αυτό ή προσπαθήσει να παρακάμψει ένα κομμάτι για να γίνουν τα έργα, αυτό δεν θεωρείται επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Είναι ένα παράδειγμα που μπορώ να σας δώσω, μπορώ να σα δώσω και πάρα πολλά άλλα. Δεν υπάρχει μια πλήρης, μια συνεκτική ανάλυση των εμποδίων που μπορούν να φράξουν το δρόμο σε όσους ε, ετούνται κονδυλίων ή μπορούν ε, να, θεωρηθούν τελικοί δικαιούχοι ετούντε. Πώς ε, αξιολογούν όλη αυτή την κατάσταση τα δύο-τρία τελευταία χρόνια, οι δικαιούχοι, οι ετούντε, οι υποψήφοι. Είπατε επίσης ε, πόσο σημαντικό είναι για τα διαφορετικά ταμεία το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και συμφωνώ απόλυτα. Το ερώτημα όμω είναι το εξή. Δεν θα πρέπει αυτό το πλαίσιο να έχει το ρόλο της δημιουργίας μηχανισμών και εργαλείων που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020. Για μένα αυτό είναι ο ρόλος ή πρέπει να είναι ο ρόλος του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσον αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιες ε, κύριες δραστηριότητες, κύριες δράσεις που θα πρέπει να αποκρίνονται στις ανάγκες ε, των μεμονωμένων περιφερειών και δαφών. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της απασχόλησης και της ε, ανάπτυξης. Υπάρχει ένα άρθρο που μιλάει για κάποια κατώτατα επίπεδα μερίδια και αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να αφορούν, να αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες των περιοχών. Τέλος. Νομίζω ότι τα εθνικά σχέδια, τα εθνικά μεταρρυθμιστικά σχέδια είναι καλύτερο σημείο αναφοράς για την πολιτική συνοχής παρά οι μεμονωμένες συστάσεις ε, για τις χώρες. Γιατί δεν ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες των κρατών μελών, που αλλάζουν συν το χρόνο. Ευχαριστώ η Μαρία Ριγκόγεν. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω το, την πρόεδρο, να ευχαριστήσω και τον Επιτρόπο. Έχω να κάνω μια ερώτηση που έχει να κάνει με το σήμερα και συγκεκριμένα με την παρουσία σας στις 16 ε, Μαΐου στη χώρα μας, στο Φόρμ για την Ευρώπη. Εκεί γίνατε ιδιαίτερα δημοφιλής ε, προς τα μέσα ε, ενημέρωσης και φέρατε πολλές ειδήσει. Είπατε ότι θα δοθεί 1,1 δις για την ανηλική απασχόληση η νεολαία μας έχει μπροστά της ένα βέβαιο σκοτεινό μέλλον και χρειάζεται σίγουρα αυτούς τους σπόρους. Όπως είπε και ο συνάδελφος Λάμπερτ, εμείς ξέρουμε πού πρέπει να είμαστε. Και ουσιαστικά το κοινωνικό ταμείο γίνεται ο κεντρικός μοχλός αυτής της προσπάθειας. Μετά λοιπόν ε, την άφηξε στη χώρα μου το Φεβρουάριο των εμπειρογνωμόνων που ήρθαν και συνεργάστηκαν με, τους, ε, με τις Ισπανικές Αρχές για να δουν πώς μπορεί να βελτιωθεί η χρήση των ταμείων και συγκεκριμένα του Κοινωνικού Ταμείου. Τι έχετε να μας πείτε και δεύτερον, ε, δεύτερο ερώτημα. Είπατε ότι θα δοθούν μάλλον άλλα 100-150 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση πάλι της νεανικής απασχόλησης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες κοινωνικής οικονομίας, οι συνεταιρισμοί μέχρι στιγμή δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση. Και ούτε έχουν απελευθερωθεί, έχουν αποδεσμευθεί κονδύλια. Ή δώσατε λοιπόν με καλές ειδήσει, αλλά ε, θέλω να μας πείτε στην πράξη ισχύουν όλα αυτά για να δημιουργηθούν ε, νέες θέσεις εργασίας για τους νέους ιδίω. Μάτουλα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά τα οποία υπόθηκαν και προηγουμένω. Μάλλον δεν θα επαναλάβω, απλώς να σας πω το εξής. Στα ευρωπαϊκά όργανα Πολλής λόγος γίνεται για υποστηρικτικά μέτρα, πολλής λόγος γίνεται για απλούστευση και ταυτόχρονη στήριξη ε, περιοχών οι οποίες ε, έχουν ε, προβλήματα, απλούστευση δηλαδή στη χρήση του Ταμείου Συνοχής κτλ δεν έχουμε ακόμα περάσει την κρίση και ούτε την έχουμε αξιολογήσει ολοκληρά, ολοκληρωτικά, αλλά βλέπουμε τώρα περικοπές δαπανών, μιλάμε για ε, πολλαπλή αιρεσιμότητα κτλ. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χάσει κάποια ε, περιοχή, ενδεχομένως πόρους από το Ταμείο Συνοχής. Εν πάση περιπτώσει, πώς βλέπετε το δεσμό, κύριε Επίτροπε, ανάμεσα ε, στην σε αυτά τα οποία θα πρέπει να στηριχτούν από το Ταμείο Συνοχής ε, από τη μία και τις κυρώσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν από την άλλη. Άλλη μία ερώτηση, την οποία ανέφηξε και ένα άλλο συνάδελφος προηγουμένω, αλλά θέλουμε και περισσότερες πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες λοιπόν για το παράρτημα 2, το οποίο είναι πιο αμφιλεγόμενο. Ε, θα πρέπει να οριστούν οι λεπτομέρειες έτσι ώστε να κατανοήσουμε περί τίνο πρόκειται. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, μια πολύ σύντομη ερώτηση η οποία σχετίζεται με αυτό που είπε ο κ. Ζέλε προηγουμένως και με τον οποίο συμφωνώ απολύτως. Ερώτηση λοιπόν κύριε Επίτροπε, δεν πιστεύετε ότι έφτασε πλέον η ώρα για να εφαρμοστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για την ευελιξία. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της ευελιξίας, ε, αλλά βάλατε και κάποια ερωτηματικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ε, ε, συζητήσαμε το 6 ε, το δημοσιονομικό πλαίσιο για το 7-13 δεν ξέραμε ότι θα προκύψει η κρίση τότε μια σειρά σημαντικών εγγράφων ε, έγιναν δεκτά, ας πούμε, η στρατηγική 2020 και μια σειρά άλλων στρατηγικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τις χώρες μέλη και μέσω των διευθυντικών ταμείων. Τα λειτουργικά προγράμματα όμως όλων των χωρών δεν εστιάζονται σε αυτές τις κεντρικές δραστηριότητες ε, και επομένως η νομοθετική ευελιξία θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε, όλους, σε όλες τις χώρες μέλη να ξαναδούν λίγο το πώς θα συνδυάσουν τα χρήματα με τις δραστηριότητες. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Yeah, ε, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Τσέλερ για την υπόδειξη ότι πάντα θα πρέπει να διευκρινίζουμε ότι τα χρήματα αυτά δεν πλέουν έτσι γενικά αδέσποτα, ότι όλα έχουν κάποιο προορισμό και ότι πάντα χρειάζεται συμφωνία και των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αλλάξει η δαπάνη των κονδυλίων αυτών. Αλλά Συμφωνώ και με την τελευταία παρέμβαση ότι θα πρέπει πάντα να είμαστε ευέλικτοι και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε και να αντιδράσουμε σε νέα στοιχεία, σε νέα δεδομένα. Η προηγούμενη Επίτροπος τα έτη 2009-2010 παρουσίασε και άξισε τις προκαταρκτικές ε, πληρωμές ε, κατά 8 δισεκατομμύρια για να ανταποκριθεί σε προβλήματα ρευστότητα που είχαν παρουσιαστεί τότε και είχαμε ε, προσαρμόσει το 1 τρίτο των μέσων μας. Φυσικά χρειαζόμαστε μία κάποια ευελιξία σε κάθε πρόγραμμα, όπως χρειαζόμαστε και μία συμφωνία, συνένεση για το ποιος είναι ο απότερος στόχος. Χρειαζόμαστε όμως και την ευελιξία. Το θέμα αυτό θα παραμείνει πάντα το ίδιο. Θα πρέπει να τονώσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα, να μειώσουμε τις οικονομικές αντιφάσεις, να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα για να διασφαλίσουμε, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Στο σημείο λοιπόν αυτών θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, αλλά η στοχοθεσία παραμένει η ίδια. Και δεν υπάρχει πιο κεντρική, αν θέλετε, προσέγγιση. Αυτό που φανταζόμαστε και δικαίω προς το συμφέρον το δικό μας και προς το συμφέρον του Ευρωπαίου Φορολογούμενου. Αυτό λοιπόν που έχουμε υπόψη είναι σε ό,τι αφορά την δαπάνη των κοντιλίων να κοιτάξουμε θέματα αποδοτικότητας και μάλιστα πιο πολύ από ό,τι μέχρι τώρα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με το περιφερειακό επίπεδο. Αλλά σε ό,τι αφορά τη χρήση και την αξιοποίηση των μέσων και την ε, εξέταση της αποδοτικότητάς τους, θεωρώ ότι αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση με την περιφερειακή διάσταση, με την περιφερειακή προσέγγιση, όχι. Θεωρώ ότι αποτελεί ε, συνέχιση της πολιτικής μας. Στη δική μου λοιπόν αντίληψη, τα ταμεία, τα διευθυντικά ταμεία δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να μεταξελιχθούν σε ένα ταμείο αντιμετώπισης της κρίσης. Όχι, παραμένουν αυτό που πάντα ήταν. Ένα ταμείο που βιώσιμα αναπτύσσει τη δομή των περιφερειών με στόχο την αύξηση του βιωτικού επίπεδου των ανθρώπων. Και ένα πράγμα που μάθαμε στο παρελθόν, και αυτό το τονίζουμε, είναι ότι αναγνωρίζουμε ότι μόνο η επένδυση σε υποδομές είναι αυτή που υστερεί. Χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα επένδυσαν επαρκώς σε υποδομές, ιδιαίτερως η Ισπανία οι υπερταχίες, ας πούμε, υπάρχουν, αλλά δεν υπήρξε ανάπτυξη της οικονομικής βάσης, επένδυση στην οικονομική βάση. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλές ε, χώρες, μάλλον αυτό προσπαθήσαμε να το βελτιώσουμε σε πολλές από τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλές από τις χώρες δικαιωνόμαστε και γι' αυτό λοιπόν οι χώρες αυτές λαμβάνουν και πολύ πιο πολλά μέσα γιατί δουλεύουν και χρησιμοποιούν τα μέσα αυτά με πολύ μεγαλύτερο εύρος επενδύσεων. Ναι, υπάρχει η πρόταση για την ελάχιστη χώρηση στον τομέα των κοινωνικών ε, προτύπων ανακατηγορία ε, ε, περιφερειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι στο σημείο αυτό απαραίτητο είναι να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχει μια ελάχιστη επένδυση σε κάποιους τομείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση της ελάχιστης. Αυτή είναι η πρότασή μας. Και τώρα σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένε συστάσεις αναχώρα, δεν θεωρώ ότι και εδώ υπάρχει κάποια σημαντική αντίφαση. Και θα ήθελα αυτό να το τονίσω επ' ευκαιρία. Δεν θεωρούμε και δεν ε, δρούμε και αναλόγως. Δεν θεωρούμε ότι βάσει των αιτήσεων συστάσεων ε, θα αλλάξουν τα προγράμματα μόνιμα. Ιδιαίτερα στη φάση της αρχής θα πρέπει να γίνουν θα πρέπει να γίνουν σεβαστές αυτές οι προδιαγραφές και αν προκύψουν ε, κάποιες αλλαγές, ε, αν προκύψουν κάποιες προκλήσεις με την πάρτα του χρόνου, θα πρέπει να αντιποκριθούμε σε αυτές. Για να απαντήσω λοιπόν στον συνάδελφο, να πω ότι στο παρελθόν νομίζω ότι έχουμε επιδείξει επαρκή ευελιξία. Αλλά να σας πω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της ευελιξίας του όλα είναι δυνατά και της ευελιξίας του προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις, διατηρώντας όμως την γενική στοχοθεσία για την Ισπανία εν συντομία. Αυτό που την προηγούμενη εβδομάδα συμφώνησε με την Ισπανική κυβέρνηση ήταν μια συμφωνία σε ό,τι αφορά τα ταμεία συνοχής για τα έτη 2000-2006 και το κλείσιμο των ταμείων αυτών προκειμένου να μπορέσουμε πιο γρήγορα να διαθέσουμε ρευστό στην Ισπανία. Να σας πω ότι η μεγάλη πρόκληση είναι τα χρήματα αυτά να μην συνδεθούν με τα ταμεία συνοχής, αλλά στις συζητήσεις μου με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών διευκρίνησα ότι θα επιθυμούσα όχι εγώ ως Επιτροπός Χαν, αλλά ότι γενικά υπάρχει επιθυμία τα μέσα αυτά να δοθούν μέσω των φροντικών ταμείων, αλλά δεν υπάρχει νομική δέσμευση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις του Μπαρόζο με την ε, κυβέρνηση την Ισπανική το ποσό είναι μεταξύ των 900 δισεκατομμυρίων και ενός 3. Και ελπίζω σύντομα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν, να τροποποιηθούν τα προγράμματα. Η μακροοικονομική διάσταση. Νομίζω ότι το θέμα της ποιότητας της ε, φοροσυλλογής ε, είναι ενδιαφέρον, γιατί όταν ε, πραγματοποιώ επενδύσεις. Σημαντικό είναι να ξέρω και πόσο βιώσιμες είναι. Και πόσο είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος για την, τον κρατικό μηχανισμό. Και αυτό θα επηρεάσει την πολιτική μας σε κάποιο βαθμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μείνουν λίγο ακόμα οι διερμηνείς, Δέκα δευτερόλεπτα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σε ξεπερίπου περίπου εβδομάδες θα ψηφίσουμε την εντολή προς τους ε, εισηγητές μας που θα ξεκινήσουν τις οργανικές διαπραγματεύσεις από τα σχόλια των συναδέλφων ε, τον τελευταίο χρόνο περίπου ή δύο, τα, τα δύο τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ποια είναι τα σημαντικά θέματα για τις διαπραγματεύσεις. Ξέρουμε που είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, που υπάρχουν αποκλήσεις. Βέβαια, στόχος είναι κοινό, η καλύτερη δυνατή πολιτική για την ανάπτυξη. Ίσως στα μέσα, στα εργαλεία διαφέρουμε, διαφοροποιούνται απόψεις μας. Πάντως ελπίζω να έχουμε καλές διαπραγματεύσεις. Αν δεν σας δούμε πριν να σας εύχομαι καλές καλοκαιρινές διακοπές, ελπίζω να μπορέσετε να ξεκουραστείτε λίγο, να κλείσει και η Κομισιόν και θα τα πούμε μετά το καλοκαίρι. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι και πολύ συχνά θα τα πούμε πριν το καλοκαίρι, αν και όχι σε αυτό το επίσημο πλαίσιο. Πρόεδρος, λοιπόν, εδώ διακόπτω και συνεδριάζουμε εκ νέου στις 3.